αναγνώρισε τα ουσιαστικά σημεία. Πραγματικά αξίζει ε, θαυμασμό. Αλλά να πω και στο Συμβούλιο πως ε, εντάξει δεν ελπίζαμε πια ότι θα γίνει τίποτα στην πρώτη ανάγνωση. Εντάξει γιατί είναι και δύσκολη υπόθεση γι' αυτό τόσο και πιο πολύ ευχαριστώ την Κομισιόν για το ότι καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση και έχουμε κάποια δυνατότητα στην δεύτερη ανάγνωση να εγκρίνουμε έναν καλό κανονισμό. Επί της ουσίας να συμπληρώσω ένα πράγμα. Κατά τα λοιπά συμφωνώ πλήρω με την εισηγήτρια και τους προλαλήσαντες. Θεωρώ όμως πως πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει εδώ πέρα η δυνατότητα καινοτομία στον κλάδο. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Σε πολλά σημεία, αν δει την Ευρώπη και το θέμα βεβαίως οπωσδήποτε της ασφάλειας, προδιαγραφές ασφάλειας υψηλές, πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Πέρα από τα, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος και αν δείτε παραδείγματο χάρη τι έγινε με το σεισμό στη Νέα Ζηλανδία και τα επίπεδα ασφαλείας που έχουμε εδώ πέρα στην Ευρώπη, βλέπετε ακριβώς το τι μας προσφέρει ε, η ενιαία αγορά. Γιατί νομίζω πως ε, τα δικά μας τα οικοδομήματα εδώ πέρα σε ένα τέτοιο σεισμό δεν θα υπέφεραν τόσο πολύ. Αλλά ταυτόχρονα βεβαίως ε, θα πρέπει να ανοίξει η κοινή αγορά για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών. Νομίζω λοιπόν πως θα επιδείχουμε έναν καλό συμβιβασμό και θα εγκρίνουμε εγκαίρως στη δεύτερη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ακούσαμε τους σκιώδεις ηγητές. Έχω και εγώ θα τα κάνω στο τέλος όμως κάποια σχόλια εκ μέρους της ομάδας. Πάντως και εμείς γενικώ συμφωνούμε με τη θέση της κυρίας Στάιλερ. Θα ακούσουμε την κυρία Βάισκερμπερ και μετά τον κύριο Σφαμπ. Δεν ξέρω αν θέλει και άλλος κανείς το λόγο. Κυρία Βάισγκερμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και εγώ δεν είμαι και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη όταν εργάζεται τόσο λεπτομερώς ε, μια συνάλφος γιατί βεβαίως έτσι αυτό αποτελεί καλή βάση, βάση της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Είναι τεχνικό και δύσκολο το θέμα αλλά μπορώ να σας πω πως παρά το ότι δεν είμαι σκιώδης ή συγγήτρια, συνεργάστηκα με τον κύριο Μάιερ γιατί με ενδιαφέρει απλά το θέμα και θα αφιερώσω χρόνο. Και αν ε, κατατεθούν τροπολογίες μην απορρίσετε, γι' αυτό είναι και τόσο λεπτομερείς οι παρατηρήσεις μου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν για τον ορισμό της κοινή θέση. Εγώ θεωρώ πως ε, επί της αρχής πρέπει να το χαιρετήσουμε. Είναι σημαντικές οι βελτιώσεις σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά τη διαφάνεια και την δεσμευτικότητα του σήματος CEE e και ενισχύεται έτσι η εμπιστοσύνη στο σύστημα συνολικά γιατί το CEE e έχει καταντήσει να σημαίνει China Export <laughs> Οπότε θα πρέπει να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το σήμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες ε, που θα πρέπει να βελτιωθούν, θεωρώ, στη δεύτερη ανάγνωση. Θεωρώ λοιπόν πως η βασική πρόθεση εδώ πέρα είναι να οδηγηθούμε σε μια πραγματική εσωτερική αγορά στα οικοδομικά υλικά, όμως, όπως λέει και η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να παραμένουν αρμόδια και οι κατασκευαστές οι ίδιοι για την ασφάλεια του προϊόντος. Και βεβαίως πρέπει να έχουν και την ευθύνη γι' αυτό. Παρά το ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προδιαγραφές ασφαλείας, ε, παραμένουν οι κατασκευαστές υπεύθυνοι. Θεωρώ επίσης πως ε, στην κοινή θέση δεν ε, υπάρχει ακόμα σαφήνεια στους όρους που μιλάει για τις ε, δηλώσεις ε, επιδόσεων ε, και εκεί πέρα δεν υπάρχουν ορισμοί για το ποια είναι η μαζική παραγωγή, ποια είναι η παραδοσιακή παραγωγή, ποια είναι η ειδική παραγγελία. Όλα αυτά είναι όροι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν ε, οριστεί εδώ μέσα, οπότε θα έχουμε πάλι διαφορετική ερμηνεία στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο βεβαίως δεν θέλουμε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ερμηνείας, αλλά αυτά τα πράγματα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή, πρέπει να είναι καλύτεροι ορισμοί. Κατόπιν, το επόμενο θέμα είναι κάπως δύσκολο για μένα γιατί εγώ είμαι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το είπε και ο πρόεδρος. Παρόλα αυτά θεωρώ πως στη δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να δούμε τις ειδικέ διατάξεις για τις μικρές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής η πρόταση της Κομισιόν εξετάζει και προβλέπει την εξέταση αυτή του συστήματος και υπάρχουν και ε, μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στην πλευρά του χρήστη. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις εγγυήσεις, γιατί εδώ πέρα εξαιρούνται πάρα πολύ από τις εγγυήσεις ασφάλειας. Εντάξει, χρειαζόμαστε εξαιρέσει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που παράγουν αυτά τα προϊόντα, αλλά όπως λέτε είναι πάρα πολλές και μικρές επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν. Και αν δεν ισχύουν οι ίδιες απαιτήσει για την ασφάλεια, ε, τότε είναι προβληματική η κατάσταση για, την, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πλευρά του χρήστη. Οπότε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι παραγωγή δεν χρειάζονται εξαιρέσεις, χρειάζονται απλούς κανόνες, αλλά όχι άλλες εξαιρέσεις προτελευταίο σημείο, ανακύκλωση οικοδομικών υλικών, γιατί αναφέρθηκε από την εισηγήτρια. Το Συμβούλιο περιορίζει στο παράρτημα 1.7 την δυνατότητα ανακύκλωσης. Τώρα το να προτιμηθεί η ανακύκλωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μία επιλογή, αλλά υπάρχει άλλη μία επιλογή, είναι η άμεση επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση. Γιατί το να ανακυκλώνονται τα υλικά δεν είναι μια φορά, ειδικά τα οικοδομικά υλικά τόσο αηφόρο. Τελευταίο επίσης σημείο για το σχέδιο έκθεσης, ε, υπάρχει μόνο στα αγγλικά αυτή τη στιγμή. Ίσως ε, να βρω και άλλες παρατηρήσεις αν μπούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά κάτι πρόσεξα είδω. Στο παράρτημα 3 μιλάτε για επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με το REACH, η τροπολογία 49. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα εδώ πέρα δεύτερη ρύθμιση πάνω από το REACH. Αν μια ουσία περιέχεται στον κατάλογο, περιέχεται. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε και σε αυτήν εδώ την οδηγία. Νομίζω πως μπορούμε να διαγράψουμε λοιπόν αυτό εδώ το παράρτημα εφόσον προβλέπετε στο ΡΙΤΣ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και χαίρομαι για την καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε κυρία Βάις Γκέρμπερ. Πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας. Ο κύριος Σουάβο, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές. Λογικό μου φαίνεται το πρόγραμμα. Δύο-τρία σημεία θέλω και εγώ σε δύο-τρία σημεία να καταθέσω τροπολογίες. Δεν αφορούν τις λεπτομέρειες, απλά για να ξέρετε πώς η ψηφοφορία μπορεί να διαφέρει κάπου από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί με το Συμβούλιο. Αλλά αυτά και τελείως ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? Έχω και εγώ κάποια σχόλια, δεν θέλει άλλο το λόγο. Και τώρα μιλώ εδώ ως εκπρόσωπος της ομάδας μου Χαίρομαι για την προσέγγιση που ακολουθεί η συγκεκριά Στάιλερ και σίγουρα υπάρχουν αισθητέ βελτιώσει, ιδιαίτερα για τι ε, μικρέ επιχειρήσει. Νομίζω ότι η συμβαστική λύση είναι πολύ θετική. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπε και η κυρία Βάι Κέρμπερ. Γίνεται διάκριση μεταξύ του γεγονό ότι οι χώρε μέλη είναι απολύτω αρμόδιε για το περιβάλλον και την ασφάλεια, για τα, τις προδιαγραφές δόμησης, ε, αντισυσμικής προστασίας κτλ. Αυτό αποτελούν απόλυτη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με το γεγονός ότι ορισμένες χώρες ζητούν ξεχωριστούς ελέγχους για τις προδιαγραφές των ίδιων δομικών ε, προϊόντων. Οπότε θα πρέπει να δούμε και τι έχουμε ζητήσει σε ό,τι αφορά το πακέτο για τα εμπορεύματα. Γιατί με το πακέτο αυτό άνοιξε η ροή πληροφοριών μεταξύ παρόχων που θέλουν να, προσχω... εισέλθουν στην αγορά και αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ερμηνείας ό,τι αφορά την νομοθεσία. Επίσης, ε, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Βάης Γκέρμπερ ότι αυτή η διατύπωση, αυτή η διάταξη για την ε, ε κοινοποίηση ε, είναι συμβατή με τις διατάξεις του ΡΙΤΣ και την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία συνεπή και συνεκτική προσέγγιση σε αυτό το σημαντικό θέμα των επικίνδυνων και χημικών ουσιών και να μην δημιουργήσουμε ξεχωριστό καθεστώς, ειδικό καθεστώς για τα προϊόντα των δομικών κατασκευών σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, ουσιών που χρησιμοποιούνται σε άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά ήταν τα δικά μου σχόλια και θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να συνοψίσει, αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε και εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωπο του Συμβουλίου, για να δούμε τι πρόοδο έχει συντελεστεί στην αρμόδια ομάδα εργασία. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Βατέσα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ θερμά και την κυρία Στάιλερ για τη σύνοψη που έκανε των βασικών σημείων και ευχαριστώ και τους σκιώδης ηγητές φυσικά που υπογράμμισαν τα πιο σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να κάνω μερικές διευκρινήσεις για αυτά που ακούσαμε. Όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά, χρειαζόμαστε μη, ένα σήμα σε ε, ε, ώστε να είναι πιο αυστηρή η ετικετοθεσία για την κυκλοφορία των προϊόντων, την εμπορία των προϊόντων. Αυτό είναι ένας περιορισμός για τις επιχειρήσεις. Φάνηκε αυτό από τις διάφορες εξαιρέσεις που θεσπίστηκαν. Στο άρθρο 5 μια στιγμή θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω τους συναδέλφους όταν πηγαίνουν έρχονται, ειδικά όταν μπαίνουν στην αίθουσα για τις ψηφοφορίες, ε, να μην κάνω φασαρία, γιατί είναι πολύ σημαντική η δήλωση του Συμβουλίου και θα ήθελα να μπορέσουμε να την ακούσουμε. Συνεχίστε. Ευχαριστώ. Στο άρθρο 5, λοιπόν, διευκρινίσαμε τις διάφορες εξαιρέσεις που επιτρέπουν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απαλλάσσονται από ορισμένου περιορισμούς του σήματο σε ε. Ιδιαίτερα για τους παραγωγούς που έχουν παραγγελία για συγκεκριμένο εργοτάξιο, για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν στο εργοτάξιο αυτό και για τα εργοτάξια που έχουν ιστορική αξία και τα συναφή προϊόντα. Τρεις είναι οι περιπτώσεις εξαιρέσεων, οπότε οποιοδήποτε μέτρο που είναι υποχρέωση για τη διαδικασία σήματος βαίνεις βάρος του ενδιαφερόμενου. Και αυτό ισχύει ουσιαστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές πλήττονται κυρίως από το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα. Επισημάνεται την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια και η υγεία υγιεινή. Είναι κοινό μας στόχος αυτός με μια μικρή διαφορά στον τρόπο ερμηνείας. Γιατί έχουμε ένα κανονισμό που αφορά τα προϊόντα. Όταν ε, μιλάτε για την εφαρμογή, φυσικά θα πρέπει εκ των προτέρων να χορηγούνται οι πληροφορίες, αλλά οι κανόνες εφαρμογής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως είπαμε, είναι κάτι που δεν αφορά τα προϊόντα, αλλά την δραστηριότητα την ε, της δόμησης. Οπότε εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για να περιορίσουμε τα ατυχήματα, γιατί περισσότερο για ατυχήματα μιλάμε παρά για νόσους. Σε ό,τι αφορά την απλουστευμένη διαδικασία, το συζητήσαμε στο Συμβούλιο, γιατί περίπου μία διετία κράτησαν οι γενικές συζητήσεις, οπότε είχαμε εκτενείς συζητήσεις για πολλά θέματα και το θέμα της απλουστευμένης διαδικασίας μας απασχόλησε αρκετά. Θα σας μιλήσω για μία από τις απλουστευμένες αυτές διαδικασίες, αυτή που αφορά τις μικροεπιχειρήσεις. Στα πλαίσια των μικροεπιχειρήσεων προσφέραμε μία δυνατότητα απλούστερης διαδικασίας, πολύ πιο απλής ε, από τη διαδικασία που ισχύει για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Φυσικά εξασφαλίζοντας την ε, σταθερότητα και την ασφάλεια ε, στα κτίρια. Φυσικά υπάρχει υποχρέωση να αποδείξουν ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, γιατί υπάρχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο επιλογής των μεθόδων, ότι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουν είναι ισοδύναμοι με αυτούς που προτείνουμε γενικώς. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε άλλα σημεία γιατί βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει και όλα τα θέματα της ανακύκλωσης αλλά και άλλα θέματα μπορούν κάλλιστα να αναπτυχθούν στον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε και στη συνεδρίαση για την ενημέρωση αυτή από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Φυσικά χρειάζεται στενή συνεργασία για να καταλήξουμε σε ικανοποιητική συμφωνία. Σας ευχαριστώ και θα είστε παρόν και στο εργαστήριο που θα έχουμε 5 Οκτωβρίου για το θέμα αυτό. Θα ξαναδώσω το λόγο κύριο, στην κυρία Στάιλερ, αλλά πρώτα να ακούσουμε τον αρμόδιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Στάιλερ για το πολύ αξιόλογο έργο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο για ένα πολύ σημαντικό κλάδο, όπως είναι ο κλάδος της δόμησης. Οι συστάσεις είναι πολύ σημαντικές και θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που αφορά τα προϊόντα και την πιστοποίηση, τα είδη των προϊόντων. Φυσικά ίσως χρειάζεται να τελειοποιήσουμε τη διατύπωση, αλλά είναι πολύ θετικό αυτό το σημείο. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες ασυνέπειες, γιατί υπάρχουν ε, απλουστευμένες διαδικασίες και STD και υπάρχει και το θέμα το Declaration of Performance, της δήλωσης επιδόσεων. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα τελειοποιήσουμε. Η κυρία Τάιλερ αναφέρθηκε σε έξι κεντρικά σημεία. Αυτό που είναι λίγο προβληματικό και εκεί ίσως έχουμε πρόβλημα με κάποιες τροπολογίες το θέμα των επικίνδυνων ουσιών είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε κι εσείς. Παρόλο που το θίξετε όχι ως πρόεδρος, αλλά ω εκπρόσωπο της ομάδας σας. Μας απασχολεί εδώ το θέμα των ε, ισχυρών διατάξεων και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνέπεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη εδώ με το REACH και να επιτείνει τη γραφειοκρατία επιβαρύνοντας τον κλάδο. Θα πρέπει να αποφύγουμε την επικάλυψη και θα το προσέξουμε αυτό σε ό,τι αφορά τι επικίνδυνε ουσίες. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι το REACH καλύπτει τη χρήση των χημικών ουσιών. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη όταν εκπονούμε επιμέρους νομοθεσία για διάφορους κλάδους. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τις γενικές διατάξεις, γιατί υπάρχουν διατάξεις στο REACH που μιλούν για επικίνδυνες ουσίες και έχει γενικό χαρακτήρα. Υπάρχει φυσικά και διαδικασία καταχώρησης και οι περισσότερες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα δομικά υλικά καλύπτονται από την πρώτη προθεσμία για την καταχώρηση που λύγει τέλη Νοεμβρίου και το REACH προσφέρει δυνατότητες για περιορισμό κάποιων ουσιών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που εμπεριέχουν. Αυτά και ήθελα απλώς να επισημάνω ότι ορισμένα στοιχεία είναι πιο προβληματικά. Ευχαριστώ πολύ. Επί του τελευταίου σημείου γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί σας της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων ασχολούνται και με την διασύνδεση με το ρίτσο και θα δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συμφωνία από αυτού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ και όλους ε, όσους ε, έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Να ξαναδώσω τον λόγο στην κυρία Στάιλε Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στη συζήτηση αυτή και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτό το κεντρικό σημείο ε, του, της, των επικίνδυνων ουσιών καθώς επίσης ε, και της ε, ετικέτας Ε είναι όντως πολύ κεντρικά σημεία. Νομίζω ότι ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας ε, και ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και τον Ρόμπερτ Φρός που με βοήθησε και στην αρχική μου έκθεση και είμαστε και καλοί φίλοι ε, και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει ίσως να ξαναδούμε τα θέματα έτσι ώστε να μην υπάρχουν φράκτες ούτε μεταξύ των γειτόνων ούτε και μεταξύ των εταιριών που ασχολούνται με την κατασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στάιλερ για την ανταλλαγή απόψεων. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Καλωσορίζω τους συναδέλφους και καθυστέρησα λίγο με τις ανακοινώσεις του Προεδρού. Θα ήθελα λίγο ίση, λίγη ισχύα. Ξέρω πως κάποιοι θα φύγετε, οπότε σας παρακαλώ να βγείτε λίγο ήσυχα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω πως και γνωρίζω πως ε, εκπροσωπώ εδώ πέρα την Επιτροπή να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας στην ε, κυρία Εύλιν Γκέπχαρτ, uh, της ο σύζυγος απεβίωσε πριν από δύο εβδομάδες. Ξέρω πως πολλοί από σας το ξέρετε ήδη, απλά θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά. Οπωσδήποτε εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή μαζί της και ξέρω πως και αρκετοί από σας το έκαναν, γιατί πολλοί από μας ε, έχουν συναντήσει τον σύζυγό της, είχαμε ταξιδέψει μαζί, την στήριζε και γνωρίζω βεβαίως πως και εσείς ε, θέλατε να μεταφέρω τα συλληπιτήριά σας. Ήθελα λοιπόν να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά και βεβαίως ε, εν καιρό αφού θα πενθήσει βεβαίως τον σύζυγό της αναμένουμε την επιστροφή της αυτό ως πρώτη ανακοίνωση για τα υπόλοιπα τώρα. Πρώτα απ' όλα να σας πω πως η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Είδαμε τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν τα σχετικά και η δική μας επιτροπή μεταδίδεται συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη επιτροπή πλην αυτής των οικονομικών. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τη δουλειά μας, το οποίο μας ικανοποιεί και Νομίζω θα συμφωνήσετε. Δεύτερον, για το θέμα της τυποποίησης για το οποίο θα ψηφίσουμε και νομίζω πως ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα και έχουμε αυξήσει την σημασία του, αλλά το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου ε, οι φορείς ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ ε, διοργανώνουν μια στρογγυλή τράπεζα εδώ μέσα όπου λέγεται σημεία κλειδιά για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης και ξέρω πως ο κύριος Κόζους είναι ο μας και η κυρία Ρούλα και Μαντρε θα είναι εκεί και ε, ελπίζω να στήριξετε αυτή την εκδήλωση. Επίσης να σας πω πως μετά τη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου στις 6 και στο σαλόνι των βουλευτών η Γενική Διεύθυνση σαν μας καλεί να γιορτάσουμε τα πέντε έτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταναλωτών που έχουμε στηρίξει. Θα λάβετε και ατομική πρόσκληση, απλά σημειώστε το, γιατί τα μέλη του δικτύου αυτού από 27 κράτη-μέλη θα είναι παρόντα, οπότε θα μπορέσετε να συναντήσετε τους εκπροσώπους σας και ελπίζω να είναι αρκετοί βουλευτές εκεί πέρα. Και τέλος να σας πω πως σήμερα το απόγευμα για το εργαστήριο για την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες, το οποίο θα διευθύνω εγώ, απουσία της κυρίας Γκέπχαρτ. Θα υπάρχει και αίθουσα ακρόασης, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζω να είστε παρόντες. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Νομίζω μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες. Ας δούμε τις ε, παρουσίες. Να ψηφίσουμε λοιπόν για να δούμε πώς είναι παρόντες. Πρώτα απ' όλα άρχεται η ψηφοφορία μόνο για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όσοι λοιπόν από το ΕΛΚ θα ψηφίσουν, παρακαλώ να ψηφίσουν τώρα. Να δούμε πώς είναι παρόντες από το ΕΛΚ. Ε, είμαστε ήδη ε, ένας παραπάνω. Μπορεί λοιπόν κάποιος να μην ψηφίσει, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα 15 άτομα. Μπορεί έλκ να μην ψηφίσει. από το ΕΛΚ να μην ψηφίσει. Ωραία, ευχαριστώ. 14 από το ΕΛΚ. Πέρας. Και μία αποχή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ψηφίσουν τώρα τα μέλη των Σοσιαλδημοκρατών, παρακαλώ. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ποιος δεν ψηφίζει. Έχουν όλες τις κάρτες τους. Ανεβαίνει σταδιακά ο αριθμός. Θέμε ώρα βλέπω. Δεν λειτουργεί η κάρτα σας. Ε, χρησιμοποιήστε ένα άλλο μηχάνημα. Απαιτείται κάποια επιτήρηση της αγοράς των καρτών, νομίζω. Λοιπόν, 10 από τους σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι. Ένα συνάδελφο έχει πάει να φέρει την κάρτα του. Είμαστε μόνο τρει. δεν με πειράζει, λέει ο πρόεδρο. Όχι, σας βλέπω εκεί, είστε τρεις, δεν χρειάζεται να ψηφίσετε οι πράσινοι. Τρεις πράσινοι σας βλέπω. Στην Ευρωπαϊκή Συντηρητική τους βλέπω. Και ψηφίζω και εγώ σήμερα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδη είναι εδώ. Όχι, είστε μόνος σας σήμερα, δεν είναι κάποιος άλλος. Ωραία. Και ο κύριος Στάς. Μπορεί να μην χρειαστούν οι κάρτες. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία για την έκθεση Κοζούσνικ. Ξέρω πως υπάρχουν πολλές συμβαστικές τροπολογίες, οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή, τον κύριο Κοζούσνικ, να κάνει μια εισαγωγή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα η έκθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος και στην Επιτροπή μας και σε άλλες επιτροπές. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν στο μέλλον. Εκτιμώ την συνεργασία μου με τους κοιόδες και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και με τις άλλες ομάδες στην ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ γιατί ήταν σημαντικό για όλους μας να γίνει αυτή η ακρόαση που έγινε κάποια στιγμή περί τα μέσα του έτους. Επίσης πήγαμε και στην Γενέβη και επισκεφτήκαμε τους διεθνούς, ε, διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την τυποποίηση. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω πως η Επιτροπή Ήτρε επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση και έχει προετοιμάσει μια δική της έκθεση και οι συστάσεις των συναδέλφων από αυτή την Επιτροπή έχουν συμπεριληφθεί εδώ πέρα. Θεωρώ λοιπόν πως έχουμε επιτύχει, δηλαδή διατηρήσαμε την εθελοντική προσέγγιση, κάτι το οποίο είναι αποδεκτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης θεωρώ πως ε, ο σκοπός όλων των εισηγητών ήταν να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοζούσνικ. Συμφωνώ. Πράγματι νομίζω πως και οι Κροάσεις και οι επισκέψεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές και έδειξε το πώς εργαζόμαστε στα θέματα της πρωτοβουλία. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με τροπολογία 12, Μπένσεν, υπέρ, κατά. Νομίζω θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία επί της πρώτης παραγράφου. Τροπολογία Μπένσον. Πέρας. Γίνεται δεκτή. 23 έναντι 13. Τροπολογία Ρούιλε 11 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 40 της Επιτροπής Βιομηχανίας με προφορική τροπολογία υπέρ κατά δεκτή. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 1 της βιομηχανίας υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 13 στην παράγραφο 3 υπέρ κατά δεκτή. Περνάμε στην 14 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά Δεκτή. Περνάμε στην 15 νομίζω κάρας ε, υπέρ κατά δεκτή ε, ήτρε δεν τίθεσε ψηφοφορία τροπολογία 16 υπέρ κατά δεκτή 17 υπέρ κατά Περνάμε τώρα συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ συμβαστική τροπολογία 1 κατά δεκτή ομόφωνα. Περνάμε λοιπόν στην 25 με προφορική τροπολογία πάλι που βλέπετε στον κατάλογο σας υπέρ της 25 κατά δεκτή. Περνάμε στην 26 υπέρ κατά Δεκτή. 27 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 32 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά Δεκτή. Ή θέλετε να επαληθεύσουμε. Ας επαληθεύσουμε. Για να μην κοιμηθείτε κιόλα. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 32. Πέρας. Δεκτή 21 με 15. Περνάμε στην 33 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. 35 υπέρ κατά απορρίπτεται 34 υπέρ θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά νομίζω 34 άρχεται η ψηφοφορία κάποιος ναι πέρας κάποιος δεν ψήφισε απορρίπτεται με 20 κατά 7 της βιομηχανίας υπέρ. Κατά. Δεκτή. Παράγραφος 10. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 39 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε λοιπόν στη συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 4 της βιομηχανίας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε. 41. Λοιπόν, άρχιτη η ψηφοφορία. Πέρασε. 26 έναντι 10 δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Δεκτή επίσης. Περνάμε λοιπόν στην 44 σε δύο μέρες. Χωριστή ψηφοφορία. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο το που είναι ο διαχωρισμός. Μέρος πρώτο λοιπόν υπέρ. Κατά. Δεκτό. Μέρος δεύτερον, υπέρ. Μάλλον θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο μέρος. αρχή την ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή με 22 έναντι 14. Περνάμε στην 45 υπέρ. Κατά δεκτή. 46 υπέρ. Κατά δεκτή. Ήτρε 14 υπέρ, κατά δεκτή. 48 υπέρ, κατά δεκτή επίσης. 47 που είναι προσθήκη στην 48 υπέρ. Νομίζω θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 47 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας 37 Απορρίπτεται λοιπόν 19 έναντι 17. Περνάμε λοιπόν στην παραγραφό 15, συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική 5 στην παράγραφο 16 υπέρ κατά και αυτή δεκτή συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά Δεκτή επίσης. Πάμε τώρα στην τροπολογία 76. Στην παράγραφο 19α νέα υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στη συμβαστική 8 λοιπόν υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 80 με προφορική τροπολογία όπως αναγράφεται στον κατάλογο υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά η τροπολογία 80 άρχεται η ψηφοφορία επί της 80 πέρας δεκτή με 33 έναντι 4 Περνάμε τώρα στην 81 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στη συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Δεκτή επίσης. Περνάμε τώρα στην 87 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 88 υπέρ. Κατά δεκτή. Περνάμε τώρα στην 9 της βιομηχανίας που είναι προσθήκη. Αυτή η προσθήκη που βλέπετε υπέρ. Κατά δεκτή. Η 89 έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία του κυρίου Μπένσον είναι προσθήκη 90 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πάμε λοιπόν στην 94. Καλά δεν λέω. Ναι, αμπάντ, σουλή, υπέρ. Κατά. Δεκτή. 95 κάποιες επιπλέον λέξεις υπέρ κατά δεκτή άρα η επόμενη δεν ψηφίζεται και περνάμε στην 16 της βιομηχανίας υπέρ κατά δεκτή Βιομηχανία 41 υπέρ κατά δεκτή 15 της βιομηχανίας υπέρ κατά δεκτή 96 Κρόιτσμαν υπέρ κατά απορρίπτεται 97 υπέρ νομίζω πως θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 97 ρέπο Άρχιε τη ψηφοφορία πέρας με μία ψήφο διαφορά 98 De Jong υπέρ κατά απορρίπτεται παραγραφούς 25 τροπολογία 100 υπέρ κατά δεκτή οπότε περνάμε στην τροπολογία 18 προσθήκη υπέρ κατά δεκτή μετά έχουμε την 101 υπέρ κατά δεκτή 102 υπέρ κατά δεκτή 103 υπέρ κατά τροπολογία 6 της ΙΤΡΕ ως προσθήκη ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΤΡΕ 42 με προφορική τροπολογία του εισηγητού ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Ήτρε 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 109. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19 ως προσθήκη της Επιτροπής Ήτρε. Κατά. Εγκρίνεται. 110. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Βλέπετε που χωρίζουν τα τμήματα. Ε, την παράγραφο 3 την έχει αποσύρει ο εισηγητής, δεν ξέρω αν την επανέφερα κάποιο άλλο μέλος. Καλώς, ψηφίσουμε χωρίς τα τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ. Α, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Στην τροπολογία 110, δεύτερο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και 15 κατά. Και το τμήμα 3 έχει αποσυρθεί. Το τμήμα 2 της Επιτροπής Ήτρε καταπίπτει. Ήτρε 22 τώρα. Ψηφίζουμε τροπολογία 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 28. 111 κρότσμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 112 ροσφόρ, ως προσθήκη, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε 35, αλλά δεν θα την ψηφίσουμε. Ήτρε 37, ως προσθήκη, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Για την τροπολογία 113, η κυρία Ρούιλε θέλει να καταθέσει και προφορική τροπολογία. Ναι, θέλω διαγραφή του όρου fundamental, θεμελιώδης, τίποτα άλλο. Στο 28α. Εκεί που λέει όταν τα φόρα και οι όμιλοι διαδραματίζουν ρόλο, όχι θεμελιώδη ρόλο. Συμφωνεί και ο εισηγητής, οπότε ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 113 με την αλλαγή κατά, εγκρίνεται. Ήτρε 27, Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ήτρε 36, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ήτρε 34, με τροπολογία στο συγκεκριμένου, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε 33, ποιος είναι υπέρ, με αλλαγές στο συγκεκριμένου, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 28F. Ήτρε 28. Ποιος είναι υπέρ με προφορική τροπολογία. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 29 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30 από τις Ήτρε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31 της Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 29. Τροπολογία 115. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 115. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 15 κατά. 115 εγκρίνεται. 116 προσθήκη του κυρίου De Jong. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69. Βερνιό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 118 με προφορική τροπολογία. Κοζουσνικ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38 τη Ήτρε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ήτρε 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 4 στις αιτιολογικές σκέψεις. Ποιος είναι υπέρ της 4 κατά εγκρίνεται. 5 και 6 πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 7 De Jong ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 ρίλε, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 με προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τελευταίες ψηφοφοριε ψηφοφορίες. 1, 2, 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνονται τα θεωρώντας. Ψηφίσαμε τις τροπολογίες. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία της έκθεσης Κόζοσνικ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια θερμά κύριε Κόζοσνικ. Πολύ αξιόλογο το έργο σας. Ελπίζουμε να περιληφθεί στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, αλλά μάλλον θα πάει για τον Νοέμβριο. Δυστυχώς, με βάση τους κανόνες του Κοινοβουλίου, δεν δικαιούνται οι σκιώδεις ηγητές χρονοαγόρευσης. Μπορείτε όμως, αν είστε στην αίθουσα της Ολομέλειας, όταν παρουσιάσει την έκθεση του κ. Κόζουσνικ, να μιλήσετε στη διαδικασία Catch the Eye. Καλό θα ήταν να είστε παρόντες. Θα ήταν θετικό και για την Επιτροπή μας και για τον κύριο Κόζουσνικ να έχουμε σημαντική παρουσία στην Ολομέλεια την ώρα της παρουσίας αυτού του θέματος. Εγώ θα είμαι πάντως. Σας ευχαριστώ και θερμά ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνατε όλοι για αυτή τη σημαντική έκθεση. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα. Έκθεση Κορέα Δεκάμπος, γνωμοδότηση μάλλον Κορέα Δεκάμπος, που θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, Πρόκειται για μια γνωμοδότηση με θέμα τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Παρακαλώ όσοι φεύγουν από την αίθουσα να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε και δουλειές. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα έχει θέμα τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ. Θα δώσω το λόγο στον ε, συντάκτη γνωμοδότηση, τον καθηγητή Φερνάντο Κορέα Campos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση, η γνωμοδότηση αυτή ε, έφτασε μια κακή συγκυρία. Γιατί ε, για λόγους σπουδής και καθυστερημένης υποβολής δεν μπόρεσαμε να λάβουμε υπόψη τη δεύτερη εκδοχή της έκθεσης Υπάρχουν πολλές διαφορές και κρεμότητες στην έκθεση. Έγιναν πολλές προσπάθειες στην λίστα ψηφοφορίας, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά θέμα εναρμόνισης ε, συντελεστών ΦΠΑ. Δυστυχώς δεν καταλήξαμε συμφωνίες σε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για την εναρμόνιση των τελεστών ΦΠΑ, παρόλο που είναι σημαντικό θέμα για το Διεθνέ εμπόριο, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθούν πολύ σημαντικά τμήματα τη γνωμοδότηση. Και θα ήθελα το λόγο πριν την τελική ψηφοφορία μου ξαναδώσατε την ευκαιρία για να εξηγήσω τη θέση μου ως συντάκτη γνωμοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους, κυρίως τους σκιώδης ηγητές, για τις προσπάθειες τους, γιατί ακόμη και με τη διαφωνία μπορεί κανείς να διδαχθεί πολύ σημαντικά πράγματα. Well, thank you very much indeed. And I think... Ευχαριστώ. Η κυρία Λεγκρίπ, που είναι σκιώδη συγγήτρια για το ΕΛΚ, θα ήθελε πριν την ψηφοφορία να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο, γιατί το θέμα το συζητήσαμε εκτενώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης, γιατί έδειξε μεγάλο πνεύμα συνεργασίας και ήταν πολύ καλός ακροατής ε, και ους σε όλες τις συζητήσεις και με ειλικρινή, στεναρό τρόπο για τις διαπραγματεύσεις, ε, με μεγάλη εντιμότητα και ειλικρίνεια και αυτό τις έκανε πολύ ενδιαφέρουσες και από ανθρώπινη άποψη. Όπως είπε και ο συγητής, ε, η έκθεση αυτή ήρθε σε μια επίκαιρη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα και σε μια κακή συγκυρία γιατί χάρη στην ανταλλαγή απόψεων, ακόμη και στην αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ μας, μπορέσαμε να καταθέσουμε πολύ σημαντικές προτάσεις και αναλλακτικέ λύσεις και παρά τη διαφωνία που παρατηρήσαμε σε πολλά θέματα, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες για να μην πω χρόνια και στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θα συνεχίσει η συζήτηση να εμπλουτίζεται από τις διαφωνίες και τις διαφορές μας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι κατέθεσα και προφορική τροπολογία, διορθώνοντας μία λέξη στην τροπολογία μου υπαριθμό 36. Εκεί τον όρο έλεγχος τον αντικατέστησα από τον όρο επίβλεψη, επιτήρηση. Καλώς. Για την προφορική τροπολογία μου λένε εδώ στη γραμματεία ότι είναι γλωσσική τροπολογία, αφορά μόνο την γαλλική μετάφραση, δεν χρειάζεται καν να την ψηφίσουμε. Είναι μια γλωσσική διόρθωση. Περνάμε στην ψηφοφορία. Και πριν την τελική ψηφοφορία θα δώσω το λόγο και στον κύριο Κορέντι Κάμπος και στην κυρία Λεκρούπ αν θέλουν ε, να κάνουν δηλώσεις. Τροπολογία είναι στην παράγραφο 1. Επειδή υπάρχουν διαφωνίες, καλύτερα να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Καταρχήν να, ελέγξουμε πώς είναι παρόντες για την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την παράγραφο 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Νομίζω ότι περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ. Βγάλετε την κάρτα σας παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 υπέρ 15 κατά. Παράγραφος 2. Άρχεται ψηφοφορία για την παράγραφο 2. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 24 ψήφι κατά. Παράγραφος 3. Ας κάνουμε ηλεκτρονικές όλες τις ψηφοφορίες. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 3. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 23 κατά. Παράγραφος 4. De Jong. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, πιο γρήγορα ψηφίζετε. Τέλος ψηφοφορίας. 14 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Για διαγραφή. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 22 υπέρ 15 κατά. Η 6 καταπίπτει. Τροπολογία 7. De Jong. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. Παράγραφος 9. Παράγραφος 6 μάλλον, τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ, 15 κατά. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της 8, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο τμήμα έχει καταπέσει. 8 δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37-19. 10. Δεκάμπος. Υπέρ. Εγκρίνεται. Νομίζω με μεγάλη πλειοψηφία. Θέλετε να συνεχίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος πάντων. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Τροπολογία 12 λοιπόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 13. Πέρας. 19 υπέρ 18 κατά. Τροπολογία 14 Κρόιτσμαν. Τι θα κάνουμε ηλεκτρονική. Τροπολογία 14 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του κυρίου Κρότσμαν πάλι. Υπέρ. Κατά. Σαφέστατα εγκρίνεται. Τροπολογία 16 του ιδίου. Υπέρ. Κατά. Ε, ε, απορρίπτεται σαφέστατα. Τροπολογία 17 του κυρίου Δεκάμπος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 18. Είναι διαγραφής. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 18. Πέρασε. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ 14 κατά, επομένως η τροπολογία 19 καταπίπτει. Τροπολογία 20 του κυρίου Κρότσμαν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται, επαναλαμβάνω. Τροπολογία 21 του κ. Δεκάμπος. Άρχεται η ψηφοφορία επί του 21, επί της τροπολογίας 21. Η 20 απερίφθη, επομένως πρέπει να ψηφίσουμε την 21. Πέρα της ψηφοφορίας ε, Απορρίπτεται. 14 ψήφοι υπέρ 23 κατά. Επομένως περνάμε στην τροπολογία 22 του κυρίου Κρόιτσμπεργκ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 Κρόιτσμπεργκ υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. Και επομένως, περνάμε στην τροπολογία 23 του κυρίου Ντεκάμπος υπέρ. Κατά νομίζω ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 23. Πέρας. Απερίφθη με διαφορά μίας ψήφου, 17 υπέρ 18 κατά. Τροπολογία 25 Κρόιτσμπεργκ υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 Κρόιτσμαν υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27, κάμφα, υπέρ. Νομίζω ότι καλύτερα να ελέγξουμε. Τροπολογία 27, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 18 κατά. Γιατί υπήρχε και μία αποχή. Τροπολογία 29 επί της παραγράφου 12. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 29 επί της παραγράφου 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ 14 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 28 Ισχύει, ναι. τροπολογία 28 λοιπόν, ως προσθήκη, άρχεται η ψηφοφορία επί της 28. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 14 ψήφοι υπέρ, 23 κατά. Τροπολογίες 30 και 31 είναι τροπολογίες διαγραφής. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τις 30 και 31. Πέρας της ψηφοφορίας. Είναι πολύ στενό το αποτέλεσμα, 18 υπέρ 18 κατά και επομένως καταπίπτει. Τροπολογία 32. Νομίζω ότι και εδώ να κάνουμε άμεσα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 32 του κ. Κάμπος. Πέρας απορρίπτεται. 13 υπέρ 24 ψήφοι κατά απορρίπτεται. Τροπολογίες 33 και 34, ε, πρόταση διαγραφής και εδώ θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία αμέσω. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 33 και 34. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται 23 ψήφοι υπέρ 13 κατά. Τροπολογία 35 Κρόιτσμαν. Υπέρ. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 35 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ 14 κατά. Τροπολογία 36. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για την τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τώρα, πέρασε τη πληροφορία. 34 μόνο ψήφισαν αυτή τη φορά, Πάντω απερίφθη η τροπολογία 15 υπέρ 19 κατά. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 37, είμαστε στην παράγραφο 16 τώρα, ψήφι υπέρ της τροπολογίας 37, κατά εγκρίνεται. Και νομίζω δεν θα ψηφίσουμε τις 38 και 39, Ωραία. Περνάμε επομένως στην παράγραφο 18 πλέον. Πρώτα απ' όλα, τροπολογία 43 έχει αποσυρθεί αυτή. Επομένως, τροπολογία 40 καμφίν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 12 υπέρ 24 κατά. Τροπολογία 44. Μάλλον να κάνουμε και εδώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της 44. Πέρας. Εγκρίνεται 30 υπέρ 5 ε, κατά. 41. Τροπολογία 41 Κρόιτσμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 41 Κρόιτσμαν. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Δύο εποχές. Και επομένως περνάμε στο 42 πλέον. The Young Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 42 προσθήκη. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 7 ψήφοι υπέρ 26 κατά. Τροπολογία 45 από διάφορους συναδέλφους ψήφοι υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 Κρόιτσμαν υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Ε, δύο λόγια του εισηγητού. Ευχαριστώ. Παρά την ε, προφανή ισορροπία των ψηφοφοριών. Φάνηκε παρόλα αυτά ο διχασμός που επικρατεί στην Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά. Φυσικά δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου, δεν είναι τραγική η κατάσταση. Θα έχουμε παρόμοιες διαφωνίες και στο μέλλον εξαιτία ε, των διαφορετικών ιδεολογιών μας. Εγώ θα καταψηφίσω την ίδια μου την ε, γνωμοδότηση γιατί πιστεύω ότι παραμορφώθηκε σε ό,τι αφορά τα βασικά της στοιχεία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμβολή τους παρά την αρνητική θέση που θα έχω στην τελική ψηφοφορία και ευελπιστώ ότι στο μέλλον τουλάχιστον θα έχουμε ευκαιρίες ε, να συμφωνήσουμε. Βεβαίω έχετε απόλυτο δικαίωμα να κάνετε κάτι τέτοιο ως και μπορώ να κατανοήσω και τη θέση σας, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά επί, της, του συνόλου της εκθέσεως. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 18 ψήφοι υπέρ 14 κατά 5 αποχές. Ε, βεβαίως, ε, αν υπολογίσουμε μαζί τις ε, ε, ψήφους τη αποχής και της εναντίον, υπερβαίνουν τις θετικέ ψήφους. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα περίπλοκο. Εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα σε λίγο. So, um, Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Αναμένουμε την κυρία Κόρατσα She was here. All right. We just need to wait a second for Mrs. Κόρατσα Μπίλτ. Την αναμένουμε λοιπόν, την κυρία Κόρατσα Μπίλτ, την αρμόδια για αυτό το φάκελο. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Um, okay, um, let's uh, then proceed with our work. And, uh, Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. Και έχουμε άλλη μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία που σχετίζεται με μια νέα πρωτοβουλία από την Κομισιόν για την παρακολούθηση του λιανεμπορίου. Θεωρούσαμε πως είναι σημαντικός τομέας για να απασχολήσει την Επιτροπή μας κυρία Κόρα Τσαμπίλ θα είναι η συγγήτρια και σωστά νομίζω φρόντισε να μας κάνει μια παρουσίαση κομισιών και ο Ζαν Καζεβάν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Μεσοτερικής Αγοράς και φίλος της Επιτροπής μας έχει έρθει να μας τα παρουσιάσει. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα την κυρία Κόρα Τσαμπίλ αν θέλει να πει κάτι πρώτα απ' όλα συγγήτρια ή μπορεί να μιλήσει μετά την παρουσίαση. Θα την ακούσουμε λοιπόν πρώτα, μετά θα δούμε την παρουσίαση εδώ πίσω μου. Μετά θα δώσω τον λόγο στους σκιώδεις ηγητές να δω ποιος είναι εδώ τις διάφορες ομάδες. Μου είπαν ότι ο κύριος Παντσέριος είναι ε, σκιώδης από τους σοσιαλδημοκράτες, κυρία Στάιλερ, Χάρτ, εγώ είμαι εδώ για τους συντερτικούς. Ρούλα, δεν... Ε, αν μπορώ να τραβήξω λίγο την προσοχή της. Για τους πράσινους ποιος είναι εδώ για αυτή την έκθεση. Εσείς. Καλώς. Ε, έχετε, έχετε πολλή δουλειά, ναι, το ξέρω. Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ. Ωραία. Δώσω τον λόγο στην κυρία Κόρατσα και μετά θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Βεζένα. Ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν η Κομισιόν θα παρουσιάσει αυτή την εξαιρετική έκθεση. Εγώ θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή και να σας υπενθυμίσω πως δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση ή πρόταση από την Κομισιόν. Η πρόκληση είναι να δούμε στην ευρύτατη αυτή έκθεση της Κομισιόν τα προβλήματα, τους περιορισμούς, τα εμπόδια, και το τι μπορεί να γίνει για να λειτουργήσει καλύτερα η λιανική αγορά. Είναι καλή η στιγμή και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή είναι η πρώτη μου έκθεση. Η λιανική αγορά δίνει δουλειές σε 17,5 εκατομμύρια ανθρώπους και, είναι, και γύρω στο 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οπότε είναι σημαντικό για να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Θα ήθελα ως βάση να έχουμε αυτό το, την λιανική αγορά για το να ξαναξεκινήσει η αγορά σύμφωνα με την έκθεση Μόντι και θα πρέπει να εργαστούμε στο πλαίσιο της δέσμευσης της ε, Κομισιόν και της Επιτροπής μας, το εγχείρημα δηλαδή που αναλαμβάνουμε με το νέο νομοθέτημα για την ενιαία αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση, είναι μια δημιουργική διαδικασία γιατί δεν έχουμε πρόταση από την Κομισιόν και με τους ενδιαφερόμενους. Η Βελγική Προεδρία στα συμπεράσματά της ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα ασχοληθεί με την... τον νόμο περί ενιαίας αγοράς αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα προκύψει λοιπόν από αυτό το νομοθέτημα για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε και να μην είναι επικαλυπτόμαστε. Οπότε αναμένω τώρα να ακούσω την Κομισιόν. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή είναι πως δεν θέλω να περιορίσω τη συζήτηση και εγώ θα δώσω έμφαση στον τομέα της λιανικής των τροφίμων που είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του τομέα λιανικής. Αυτά και αναμένω να ακούσω τι θα πει η Κομισιόν. Ωραία. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή. Μου θύμισε ο εδώ πέρα πως πρέπει να προσέχουμε λίγο γιατί δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζητήματα τροφίμων και γεωργίας. Οπότε πρέπει να είναι σαφές πως μιλάμε για την ηλιανική, αλλά ναι βεβαίως και το τρόφιμα είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον Ζωάν Βεζεμό να λάβει τον λόγο. Εγώ θα φύγω για να μην βλέπετε το κεφάλι μου συνεχώς, θα καθίσω στην άκρη και αναμένω αυτά που έχετε να πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση στην Επιτροπή σας και συνειδητοποιώ πως ο χρόνος πιέζει και γνωρίζω πως είστε αυστηρός οπότε σας παρακαλώ εάν μακρηγορώ πείτε μου να συντομεύω. Η έκθεση αυτή ευθύθηκε στις 5 Ιουλίου και Θα διατρέξω τους στόχους στην παρουσίαση. Σκοπεύω να εξετάσω τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα τους στόχους. Δεύτερον, να εξηγήσω πως εμείς θεωρούμε πως έχουμε μια νέα καινοτόμο προσέγγιση. Είναι η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία της Κομισιόν όσον αφορά την παρακολούθηση της αγοράς και θα εξηγήσω λίγα περισσότερα πράγματα σε λίγο. Και αυτό το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ είναι τα ευρήματα, τα κυριότερα ευρήματα ανά ομάδα ενδιαφερομένων και θα ολοκληρώσω με να σας πω πού βρισκόμαστε και πού σκοπεύουμε να τι σκοπεύουμε να κάνουμε με αυτή τη δουλειά εδώ Λοιπόν, όσον αφορά τους στόχους, αναφέρεται ξεκάθαρα στην έκθεση πως αυτό το οποίο θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι θα εφαρμόζονται ελευθερίες εσωτερικής αγοράς για να διασφαλίσουμε έντονη βεβαίως οικονομική, οικονομικές επιδόσεις αλλά σεβόμενη και την εδαφική συνοχή καθώς και την προστασία καταναλωτών εργαζομένων και περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ αυτή η στόχοι αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι πως προετοιμάζοντας αυτή την έκθεση είναι πως ε, παρά το ότι το παρουσιάζει η γενική μας διεύθυνση υπήρχαν 11 άλλες γενικές διευθύνσεις, 11 συνολικά γενικές διευθύνσεις που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, μία από τις οποίες είναι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, οπότε είναι οριζόντια πρωτοβουλία και προσπαθούμε έτσι να διασφαλίσουμε πως εφαρμόζοντας τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς ακολουθούμε όλους τους στόχους πολιτικής σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται οι υπηρεσίες ε, του τομέα αυτού. Αν δείτε τον τίτλο, μιλάμε και για δίκαιες υπηρεσίες τι σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με τους στόχους του 2020 σημαίνει έξυπνες, ε, καινοτόμες, ε, προφανώς ε, αηφόρες, εκεί όπου να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το λιανικό εμπόριο και στις επιχειρήσεις στην ίδια τη λειτουργία του βεβαίως, αλλά και με το να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε διαφορετικά αποτελέσματα και όπως ανέφερε η συγγετρία Μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικό πόλο απασχόλησης ε, στο μαήθος που έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Και γιατί δίνεται αυτή η έμφαση στην ε, δικαιοσύνη. Βεβαίω ε, για να ακυρωθούν οι ακρότητες του οικονομικού φονταμεταλισμού. Βεβαίω μιλάω στους πολιτικούς, δεν θέλω να κάνω πολιτικές δηλώσεις, αλλά συχνά θεωρείται πως ε, εδώ πέρα με τη λιανική καταπολεμάμε τον πληθωρισμό και βεβαίως εντάξει είναι κάτι το σημαντικό αυτό που θα πρέπει να συνεχιστεί ειδικά στον αφορά τους καταναλωτές αλλά δεν είναι αυτό το μόνο η μόνη λειτουργία. Υπάρχει και ένας ποιοτικό ρόλος. Οι καταναλωτές δεν θα είναι μόνο φτηνά προϊόντα, θα είναι και πρόσβαση σε πολλά προϊόντα, σε ποικιλία προϊόντων και ποιοτικά προϊόντα. Οπότε, τι λέμε εδώ κατ' ουσία. Δεν πρέπει να σώσουμε μόνο τον να βλέπουμε μόνο τον τομέα της λιανικής ε, από την πλευρά του ανταγωνισμού των τιμών. Πρέπει να το δούμε από το φως όλων αυτών των πτυχών. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην έκθεση αυτή. Είναι λοιπόν μια νέα προσέγγιση για την Κομισιόν. Όπως είπα, προσπαθούμε να δούμε όλους τους στόχους μας και βεβαίως η Επιτροπή μας το αντιλαμβάνεται αυτό και εφαρμόζουμε τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς και συνεχώς ε, τίθενται ερωτήματα του τύπου πως εάν ανοίξουν περισσότερο το διασυναριακό εμπόριο πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κοινωνική προστασία, προστασία των τα κτλ. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο για εσά. αλλά πρέπει να εξηγήσουμε πως είναι καινοτόμο για εμάς και νομίζω ήταν και ικανοποιητικό να συνεργαστούμε με συναδέλφους από τις 11 άλλες γενικές διευθύνσεις έτσι ώστε και οι πολιτικές τους να ενσωματωθούν εδώ πέρα και να βρούμε τη σωστή ισορροπία που είναι πάντα αυτό το οποίο κάνουμε όταν αναπτύσσουμε πολιτικές εσωτερικής αγοράς. Επίσης, ταιριάζει με αυτά τα οποία είχε πει η έκθεση Μόντι και νομίζω πως και αυτή η λογική ενσωματώνεται εδώ πέρα. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής είναι πως δεν παραγγείλαμε πολλές μελέτες και μετά τις αντιγράψαμε. Αυτό έγινε με βάση έρευνα, έρευνες των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, συνεντεύξεις σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών, όπου οργανώθηκαν συναντήσεις μεταξύ διαφόρων υπουργείων, καθώς πολλά υπουργεία ενδιαφέρθηκαν, αλλά και με τους ενδιαφερομένους που ήταν πάρα πολλοί. Οπότε Ήταν ε, εσωτερική δουλειά αλλά και με διαβούλευση και θα δείτε πως αφενός υπάρχει η έκθεση που συνοψίζει τα κύρια ευρήματα και τη λογική της προσέγγισης αυτής και από την άλλη θα δείτε και τα έγγραφα εργασίας του προσωπικού και την έρευνα σε μεγάλο βαθμό και τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε. Επιμείναμε στο να δούμε το τι θα γίνεται και προς τα πάνω και προς τα κάτω σχέση με αυτόν τον κλάδο, δηλαδή το τι αναμένουν οι καταναλωτές, τι υπηρεσίες λαμβάνουν, αλλά και τον ρόλο του κλάδου αυτού στην διευκόλυνση του διασυναριακού εμπορίου για τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές που χρειάζονται βεβαίως στον τομέα της λιανικής για να φτάσει το προϊόν τους στην αγορά. Οπότε αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ε, επιλέξαμε τον τομέα της λιανικής για επιτήρηση της αγοράς, γιατί συνδυάζει όλους αυτούς τους συνδέσμους και βεβαίως σχετίζεται με την αγορά εργασίας, με παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, χρησιμοποιεί και ε, βασίζεται σε πάρα πολλές ε, υπηρεσίες για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Προφανώς εξετάσαμε τις διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την απόδοση του τομέα τις διαρθρωτικές οικονομικές διαφορές και τις ρυθμιστικές στον βαθμό που μπορούσαμε να διαπιστώσουμε και από αυτόν τον αρχικό έλεγχο και θα βρείτε βεβαίως στο τέλος ε, του εγγράφου έναν κατάλογο καταλήξαμε σε 20 προβλήματα θα λέγαμε της εσωτερικής αγοράς και χαίρομαι για το ότι η Επιτροπή σας αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί τώρα τι κάνουμε. Ρωτάμε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο ποιο από τα προβλήματα αυτά πρέπει να μας απασχολήσει. Όσον αφορά λοιπόν τα κύρια ευρήματα, από την πλευρά του καταναλωτή, ένα από τα βασικά ζητήματα προκύπτει είναι η έλλειψη προσβασιμότητας σε φθηνές υπηρεσίες λιανικής. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι κριτική στον τομέα της λιανικής, αλλά είναι σαφές πως αυτό είναι ζήτημα για τις ε, περιοχές της Υπέθρου, σε περιοχές του κέντρου των πόλεων, υποβαθμισμένες, η έλλειψη η μαγαζιών λιανικής σε μικρή απόσταση. Μπορώ να δεχτώ ερωτήσεις, αλλά βρήκαμε πως οι αιτίες μπορούν να είναι οι βλέπετε ε, πως υπάρχουν οι κανόνες οι πολεοδομικοί. Εγώ δεν είπα βεβαίως πως θα πρέπει να ασχοληθεί η Κομισιόν με αυτά τα ζητήματα τοπικού επίπεδου, αλλά ξέρετε πως η οδηγία για τις υπηρεσίες ε, βοήθησε να φύγουν λεγόμενες ε, οικονομικές δοκιμές λεγόμενες. Οπότε τι έγινε. Εξυγχρονίστηκαν τα κράτη-μέλη, αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε πως η λογική η οποία υπάρχει ε, εμφανίζεται στο επίπεδο της χωροταξίας, της πολεοδομίας, σύμφωνα με τα ευρήματά μας στην έκθεση. Είναι σημαντικό αυτό στη συζήτησή μας με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εάν το όφελος της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να φτάσει παντού, θα πρέπει όλα τα ε, επίπεδα και οι αρμόδιες αρχές ε, να συνεργαστούν και είναι ενδιαφέρον πως υπάρχουν διασυνοριακές διαφορές που οδηγούν ξεκάθαρα σε στρεβλώσεις. Και ε, ρωτήσετε τους αδέλφους στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής υπολογίζουν πως γύρω στο 35% των πολιτών, ένα τεράστιο νούμερο, ζουν σε μεθοριακές περιοχές. Οπότε αν υπάρχουν ε, τέτοιες ε, επιπτώσεις που διαχέονται είναι σαφώς ένα ζήτημα ιστορικής αγοράς. Μετά είδαμε πως υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες και μπορώ να σας πω πως από όταν κυκλοφόρησε αυτή η έκθεση υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και από τον τομέα της λιανικής και από αυτή την αγορά όσον αφορά τους κανόνες ε, για την ανάπτυξη νέων κέντρων κτλ. Οπότε φαίνεται πως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα και θα βρείτε κάποια πράγματα προξενούν έκπληξη όπως το ότι τα νίκια ανεβαίνουν σε κάποια νέα σε σχέση με τα παλαιότερα. Οπότε υπάρχουν σαφώς τις λειτουργίες στην αγορά. Δεύτερο σοβαρό πρόβλημα για τους επιχειρηματίες της Ελληνικής. Πέρα από το πρόβλημα εισόδου στην αγορά το οποίο, το οποίο ανέφερα, λόγω των διαφορετικών κανόνων και της ε, χωροταξίας. Υπάρχει η αγορά βεβαίως της επαγγελματικής στέχης, αλλά διαφέρουν και οι κανόνες όσον αφορά τη δικαιόχρηση που είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το τομέα και σε άλλους. Εάν θέλει κάποιος δηλαδή να αναπτύξει μια νέα μορφή επιχείρησης για να αναπτυχθεί γρήγορα, δουλεύει μέσω του franchising. Οι διαφορετικοί λοιπόν κανόνες για τη δικαιόχρηση τους εμποδίζει να το κάνουν αυτό διασυνοριακά. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τους λιανοπολιτές και θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια και τους διαφορετικούς κανόνες για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Είναι ευαίσθητο αυτό το θέμα. Σε τι αναφέρομαι εδώ πέρα. Μας είπαν οι άνθρωποι της Λιανικής πως δεν μπορούν να βρούνε προϊόντα, μάρκες από άλλα κράτη-μέλη λόγω του ότι ε, είναι, υπάρχουν περιορισμοί στην εμπορία τους. Βεβαίω αυτό αυστηρά δεν είναι αλλά είναι πρόβλημα εσωτερικής αγοράς γιατί εάν προσπαθεί κάποιος να προμηθευτεί κάτι διασυνοριακά μπορεί να υπονομεύει κάτι που είναι ε, βεβαίως στην αγορά στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς και υπάρχουν τέτοια στοιχεία στο κείμενο τώρα όσον αφορά τους προμηθευτές που βασίζονται πάρα πολύ στον τομέα αυτών. Αυτοί έχουν πρόβλημα με τους κανόνες προς μια άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή οι κανόνες περί αθέμη του ανταγωνισμού σημαίνει πως έχουν φοβερές απαιτήσει από εμάς οι λιανοπολιτές. Υπάρχουν Υπάρχει κριτική για την ίδια ετικέτα των καταστημάτων. Ε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω λοιπόν είναι πως οι κανόνες ε, που ισχύουν για να ρυθμιστούν ε, αυτά τα ζητήματα διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ των κρατών μελών και επ' αυτού του ζητήματο προφανώς συνεργαζόμαστε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, αλλά αυτό το οποίο θα έλεγα στην Επιτροπή σας είναι πως αυτά δεν αντιμετωπίζονται όλα με το δίκαιο του ανταγωνισμού Υπάρχουν ζητήματα αριθμιστικά για τον αθέμητο ανταγωνισμό και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε πώς οι... και διαπιστώνουμε πως οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ένα άλλο ζήτημα προέκυψε είναι το θέμα του υψηλού κόστους. Οι προμηθευτές θέλουν και είναι θετικοί και εδώ πέρα μιλάει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συνεργαστούν με τους λιανοπολιτές για τα προϊόντα δικής τους ετικέτας, όπου αναπτύσσουν ετικέτες ποιότητας, ειδικά όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά τι βλέπουν. Επενδύουν για να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στις ετικέτες που έχουν οι λιανοπολιτές, αλλά αν θέλουν σύμβαση με άλλον πολιτή σε άλλο κράτος μέλος δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή δεν λέω πως ε, εάν κάποιος συνεργάζεται με μία μάρκα στην Ιταλία και όχι στη, στη Γαλλία που δεν υπάρχει στην Ιταλία πρέπει να επιβάλλει το σήμα του και στην Ιταλία αλλά όταν μιλάμε για εφαρμογή προδιαγραφών, πιστοποίηση κτλ. Σημαίνει αυτό μια τεράστια επένδυση από μια μικρομεσαία επιχείρηση και το να μην μπορεί να ανακτήσει αυτή την, επιχείρηση, την επένδυση, να μην του αναγνωρίζεται όταν συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις σε άλλα κράτη-μέλη. Και αυτό βεβαίω επανέρχεται στους καταναλωτές γιατί είναι πολύ θετική για τις ποιοτικέ ετικέτες, αλλά από την άλλη παραπονιούνται πως δεν είναι καμιά φορά απολύτως σίγουροι το ότι αντιπροσωπεύουν αυτά και υπάρχει άποψη πως είναι εθνική και κατακαιρματισμένη η αγορά. Ένα σημαντικό λοιπόν ζήτημα. Τώρα, οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης, όπως είπαμε είναι τεράστιος αυτός τομέας από πλευράς απασχόλησης, είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά το πρώτο είναι το πρώτο σημείο εισόδου για ανειδίκευτους ανθρώπους και παίζει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, παρόλα αυτά. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι για την αγορά εργασίας, αλλά χαρακτηρίζεται και από πολύ μεγάλη ποικιλία, ακόμα και εντός των κρατών μελών, όσον αφορά τις συλλογικέ συμβάσεις που αφορά το κλάδο, τον τύπο, το μέγεθος εταιρείας, και αυτό μας οδηγεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την επιβολή. Δεν είναι θέμα δηλαδή του να λέμε οι κανόνες, γιατί πρώτον είναι πολύ κατακαιρματισμένος ο κλάδος, δηλαδή εμείς σκεφτόμαστε τις μεγάλες εταιρείε, αλλά είναι πολύ σημαντικό τομέα όσον αφορά τις μικρές εταιρείε και ελπίζουμε πως θα συνεχίσει να είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι πω εάν προσπαθεί κάποιος να ανταγωνιστεί με το να βελτιώσει τις συνθήκες απασχόλησης και υπάρχει μια πολύ μεγάλη άτυπη οικονομία με την οποία ανταγωνίζεται, είναι πολύ δύσκολο να βελτιώσει τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά και αυτό είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Οι οργανώσεις των καταναλωτών θα σας πούν πως κατά κανόνα υπάρχουν ηλιανοπολιτές που έχουν το καλύτερο σύστημα παραπώνων και πληροφόρησης των καταναλωτών είναι αυτές οι οποίες έχουν καλές συνθήκες εργασίας και ικανοποιημένο προσωπικό. Γιατί βεβαίως η δουλειά αυτή είναι ανθρωποκεντρική. Είναι η σημαντική απασχόληση και οι επιχειρήσεις θέλουν να το βελτιώσουν αυτό. Οπότε ο κατακρεματισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός. Όπως είπα η άτυπη οικονομία που είναι πρόβλημα βεβαίως για όλους τους τομείς υπηρεσιών, είναι πρόβλημα κλειδί εδώ πέρα και εμποδίζει την ανάπτυξη πιο ποιοτικών πρακτικών εργασίας και τη διάχυσή τους. Κάτι ενδιαφέρον, παραπονιούνται οι καταναλωτέ πω δεν ξέρουν πάρα πολλά για το τι κάνει στο κοινωνικό πεδίο ε, η επιχείρηση ηλιανική πώληση το ανέφερα και θα σα πούνε βεβαίω τις ετικέτες τους, τις ποιοτικέ, τις ηθικές κλπ που είναι πλέον κάτι το, το οποίο αναπτύσσεται και στην κρίση, δηλαδή μπορεί να μείνουν άλλα έξοδα, αλλά παραμένουν πιστοί σε αυτές τις ετικέτες. Αλλά τι γίνεται εντός του κλάδου Ξέρουμε ότι ο αγρότης, ας πούμε, είναι στην αρχή της ε, αλυσίδας, αλλά δεν ξέρουμε ότι ενδεχομένως οι συνθήκες εργασίας ενός λιανέμπορα ε, μπορεί να είναι ε, πάρα πολύ κακή. Αυτό δεν είναι κριτική προς τους ασχολούμενους με το λιανικό εμπόριο. Είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο και που παρά αυτά θέλουν να έχουν την σωστή πληροφόρηση και να κάνουν τις τις ε, τελευταίες καινοτομίες. Τελευταίο, αλλά όχι μικρή σημασία, στο θέμα των δεξιοτήτων. Όπως ε, έχω ήδη και ε, προηγουμένως, πολλοί ασχολούνται πρώτη φορά στη ζωή τους επαγγελματικά στο λιανεμπόριο, ας πούμε, από όταν είναι φοιτητέ, βρίσκουν κάποια δουλειά στο λιανικό εμπόριο. Είναι ε, πρέπει να πούμε όμως ότι το λιανικό εμπόριο είναι ο τομέας όπου όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται ε, οι η πληροφορική, χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, ε, αλλά βεβαίως χρειάζονται εργαζόμενοι με δεξιότητες που από τη μία πλευρά να γνωρίζουν τι είναι λιανικό εμπόριο και να καλύπτουν τις απαιτήσει του λιανικού εμπορίου, ενώ από την άλλη πλευρά να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι ε, κεντρικής ε, σημασίας ε, θέματα και νομίζω ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν από αυτό και αναφερόμενοι στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον κλάδο ακριβώς λένε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση και ανταπόκριση των ε, δεξιοτήτων. Ε, βλέπουμε προς το μέλλον. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μονάχα τους καταναλωτές ε, της σήμερα, αλλά και τους αυριανούς. Θέλουμε να προβλέψουμε τις, τον τρόπο συμπεριφοράς τους και επομένως το λιανικό εμπόριο θα πρέπει να εξελιχθεί με τρόπον ώστε ε, να, και τα επιχειρηματικά του προγράμματα να αναπτυχθούν με τρόπο ώστε να ανταποκριθούν στην, ε, στη μελλοντική ζήτηση και επομένως να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αηφορίας. Ε, το κόστος μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά θα καλυφθεί από την ίδια την ε, αλυσίδα των προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λιανικό εμπόριο δεν ε, μπορεί να έχει δικές του ε, στατιστικές όσον αφορά την χρήση με πούμε, ενέργεια ή την περιβαλλοντική επίπτωση. μιλάμε ο, πολλές φορές ε, λαμβάνουμε υπόψη ε, την ε, ψυχτική ας πούμε ικανότητα μιας εταιρεία την δυνατότητα να βρίσκεται σε κτίρια τα οποία έχουν καλό περιβαλλοντικό παράγοντα. Βεβαίως μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον. Μπορούμε να σκεφτούμε ενδεχομένω την ανάπτυξη των λεγόμενων green shops, πράσινων καταστημάτων και βλέπουμε ότι κάποιοι φορεί και κάποιες χώρες ε, είναι πιο θετικά διακείμενε όσον αφορά τέτοιου είδους ε, διαδικασίες. ακόμα δεν έχουμε ε, μια κοινή μεθοδολογία για τα πράσινα προϊόντα και αυτό γιατί ορισμένες ε, χώρες ε, προτρέχουν κατά κάποιο τρόπο και επιβάλλουν ήδη πράσινη μεθοδολογία για προϊόντα ενώ σε άλλες χώρες τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει τόσο. Υπάρχει μια κατάκριση. Επίσης, γίνονται διάφορες ε, μελέτες όσον αφορά τον ε, σχεδιασμό ε, της αστικής ικανότητας, δηλαδή νέους τρόπους delivery, νέους τρόπους αντιμετώπισης της ζήτησης. και εν πάση περιπτώσει είναι, ε, ε, ίσως είναι απλοϊκό αυτό που θα πω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε ας πούμε την ε, συμφόρηση στις πόλεις μας, θα ήταν πιο έξυπνο αντί να παίρνουμε εμείς αυτοκίνητό μας και να πηγαίνουμε στο μαγαζί, το μαγαζί να έρχεται σε εμά. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχει μεγάλο ε, ε, μεγάλη, ε, μεγάλο περιθώριο δυναμικής εξέλιξης το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε γενικές γραμμές εμείς βλέπουμε ότι είναι ακόμα πολύ μικρά τα ποσοστά του ηλεκτρικού εμπορίου. Υπάρχουν διάφορα βιβλία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά τελικά ε, τα ποσοστά εξακολουθούν ακόμα να είναι χαμηλά. Οι ίδιοι οι ανέμποροι θα πρέπει να ασχοληθούν, να στραφούν προς το ηλεκτρονικό ε, εμπόριο. Ναι, θα, θα τελειώσω. Μονάχα την τελευταία διαφάνεια. Είχαμε πάνω από 100 απαντήσεις. Και όπως είπε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ε, ε, προηγουμένως, ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σαν μέλος της εσωτερικής ενίας αγοράς. Στις 27 Οκτωβρίου θα έρθουμε, έχουμε μια συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και βεβαίως θα αναφερθούμε αργότερα ενώπιόν σας για το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής. Ε, τώρα, εμείς κάνουμε τη δικιά μας εργασία, θα θέλαμε να ξέρουμε και τι, τι θεωρείτε εσείς ε, προτεραιότητα, ε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε μαζί. Και βεβαίως η εργασία μας εκτείνεται οριζόντια. Ασχολούμαστε και με άλλα παρεμφερή ζητήματα, τα οποία εντάσσουμε τελικά ε, στην εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να αναφερθώ στα θέματα αυτά και περιμένω βεβαίω και τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή σας και θα ήθελα πριν ε, περάσουμε στη συζήτηση να κάνω και εγώ ένα σχόλιο διαπίστωσα ότι στην αρχή πολλές αυτές τις προτάσεις για την ε, οριζόντια προσέγγιση και την βράξη ε, ενιαίας αποδώσατε στην έκθεση Μόντι. Η δική μας επιτροπή με την έκθεση Brex ουσιαστικά είχε την ιδέα για το Single Market Act. Φαίνεται όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέχασε τελείως το ρόλο που διαδραματίσαμε εμείς δεν σας διέκοψα το, το φέρατε, αλλά ελπίζω να διαβιβάσετε στους αρμοδίους ότι της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς ότι δεν είναι μόνο ο καθηγητής Μόντι, αλλά και η δική μας επιτροπή που έθεσε το σωστό, τη σωστή βάση για αυτή τη συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγητριά μας και μετά στους Κιώδης. Λέω και Τριανταφυλλίδης, Τάιλερ, Στάιλερ θα μιλήσει για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και μετά τους σκιώδης ηγητές. θα λάβω και εγώ το λόγο ως σκιώδης. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ Μάλκολ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ευρυθή και πολύ επαγγελματική έκθεση που υπέβαλε θα μας βοηθήσει στην αναζήτηση σημαντικών λύσεων. Και εγώ είμαι μικροεπιχειρηματίας και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε πολύ εύχριστες λύσεις και αποτελεσματικές. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ορισμένα μόνο θέματα. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Το πιο σημαντικό πάντως αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρώπη. Και το λιανεμπόριο θα διαδραματίσει εδώ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης της απασχόλησης. Δεν θα απαριθμίσω τις δικές μου προτεραιότητες. Προτιμώ να ακούσω τους συναδέλφους πρώτα. Εγώ έχω αποκρισταλωμένες απόψεις για πώς θα πρέπει να χειριστούμε τις διάφορες σχέσεις εργοδοτών, εργαζομένων, καταναλωτών, διανομέων, και τα ενεργειακά θέματα, αλλά προτιμώ να ακούσω πρώτα τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτριά μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρουσίαση της έκθεσης μας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη. Δίκιο έχετε ότι το θέμα της απασχόλησης είναι κεφαλαιόδες και φυσικά η μεταχείριση των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο. Πολύ σωστά μας περιγράψατε και το μεγάλο φάσμα των διαφορών. Ορισμένοι λενέμποροι «Ε, επενδύουν ε, σε επιμόρφωση, κατάρτιση, ανάπτυξη των προσόντων, αλλά όχι όλοι. Πώς θα ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτούς που δεν επενδύουν σε τέτοια θέματα στο, που δεν επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, πώς θα τους παροτρύνουμε για να το κάνουν εκθέτοντάς τους, ξεμπροστιάζοντάς τους, κατά κάποιο τρόπο προσπαθώντας να τους κηρύσουμε το φιλότιμο, με ποιο τρόπο θα τους δώσουμε ενάψματα και πώς είναι οι λιανέμποροι που εφαρμόζουν ε, το ε, EFQM σε ό,τι αφορά την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και γνωρίζω από την προσωπική μου πείρα στην Σκοτία και τη συνεργασία μου με το αντίστοιχο συνδικάτο που εκπροσωπεί τους λιανέμπορους. Προσπαθούμε να Είχαμε σημαντική εκστρατεία κατά της βίας στον εργασιακό χώρο, πολύ σημαντική εκστρατεία, γιατί κανείς δεν θα πρέπει να εργάζεται σε έναν χώρο που υπάρχει βία. Και είναι ντροπή πραγματικά που τέτοια φαινόμενα εντοπίστηκαν και στον τομέα του λιανεμπορίου. Αν δεν είχαμε κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, δεν θα είχαμε την έγκαιρη παράδοση. Και το λιανεμπόριο βελτιώθηκε με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πριν από πολλές δεκαετίες είχαμε μεγάλη απόσταση, ε, μεγάλη πρόοδο ό,τι αφορά τις σχέσεις ε, παραγωγών, καταναλωτών, ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, νέος σχετισμός δυνάμεων στην αγορά κτλ. Συναρπαστικές εξελίξεις. Ποιο θα είναι όμως το επόμενο ποιοτικό άλμα. Μιλήσαμε για τις online πωλήσει και πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες να αγοράζουν ε, διαδικτυακά και να τους παραδίδονται στο σπίτι τα προϊόντα. Δεν έχουν όμως όλη πρόσβαση σε online αγορές. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και οι καταναλωτές ε, που διαμένουν σε απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε online αγορές. Μερικές φορές ε, είναι πολύ διαφορετικές οι οικονομικές συνθήκες και σε ορισμένες περιοχές είναι πολύ πιο αντίξωε. Και το λιανικό εμπόριο πλήττεται ιδιαίτερα από αυτές τις διαφορές. Ε, Επίση είναι και το θέμα των ακινήτων ε, που αγοράζουν ε, οι άνθρωποι και που επενδύουν η ύφεση πάντως χτύπησε όχι μόνο τον τομέα των ακινήτων και το στεγαστικό, αλλά και το ελληνικό εμπόριο. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Το ανέφερε και η συγκήτρια. Ορισμένοι λιανέμποροι προσπαθούν να περιορίσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να τις μηδενίσουν αν γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προάγουμε τι ε, βέλτιστες πρακτικέ. Πώς θα το κάνουμε όμω, γιατί έχουμε τους τέσσερις άξονες, γιατί να βάλουμε ένα πέμπτο και το περιβάλλον. Επίσης μιλήσαμε για τις χαμηλές αμοιβέ στο εμπόριο. Πολλοί εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο επιτελούν τεράστια έργο, αλλά δεν ε, επιβραβεύονται αντίστοιχα ή δεν αναγνωρίζεται η αξία τους όπως θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ πάντως για την παρουσίαση και αισθάνομαι ότι φεύγω πολύ πιο ενημερωμένη από ότι ήρθα στη συνεδρίαση για το θέμα του λιανικού εμπορίου. Ευχαριστώ, Κάθριν, ο κύριο Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έθεσε το πλαίσιο στη συζήτηση. Θα συνεχίσω στα δανέζικα. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και ο κλάδος του ελληνικού εμπορίου. Και είναι και ευρύτατος, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Και φυσικά ήταν πολλές οι γενικές διευθύνσεις που αναμίχθηκαν και ορισμένες προτάσεις του Επιτρόπου Μπαρνιέ φαίνεται ότι αλλοιώθηκαν κάπως. Έχουμε σημαντική πρόκληση ενώπιον μας θα πρέπει αυτό το ευρύτερο φάσμα να το περιορίσουμε κάπως και να είμαστε πολύ πιο επικεντρωμένοι στις δράσεις μας. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες και να πω και σε εμά να κάνουμε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να εξετάσουμε τις τεράστιες διαφορές στις τιμές που ισχύουν στην εσωτερική αγορά που αντανακλούν την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς. Επίσης το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά. Επίσης υπάρχουν θέματα ενοχικών υποχρεώσεων, πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Περιμένω με ανυπομονησία και την έκθεση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας. Εντοπίστηκαν 20 τομείς ό,τι αφορά τις σχέσεις ε, επιχειρήσεων και πολιτών. Προτιμώ να επικεντρωθούμε σε πολύ λιγότερους τομείς και να εντοπίσουμε και τους μηχανισμούς που θα χρειαστούμε στο μέλλον για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Γιατί να μην διοργανώσουμε και μια δημόσια κρόση με το θέμα αυτό, με εκπροσώπους ε, των οργανώσεων εμπόρων ή των εταιριών. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το ελληνικό εμπόριο είναι οι πλέον αρμόδιοι για να μας πούν τι χρειάζονται. Να φέρουμε σε μία μήνυα ακρόαση και εκπροσώπους φυσικά των οργανώσεων καταναλωτών και να ακούσουμε τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων. Επίσης, ε, επιμένω στο ότι θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής ε, της έκθεσης. Ελπίζω ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Πολύ καλή πρόταση. Θα τη σχολιάσει αργότερα η συγγετριά μας, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Και όπως είπε ο κύριος Μπερζεβάν, ορισμένα θέματα περιλαμβάνονται και στο European Single Act. Single Market Act. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Κυρία Ρούλε. Και εγώ συμφωνώ, ήταν όλα αυτά συναρπαστικά. Όπως σας είπα, το συζητήσαμε αυτό και στην ομάδα μας. Πρέπει να δούμε τώρα ποιος θα αναλάβει την Κοιτάξτε, το συμπέρασμά μου και εμένα είναι πως πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Δεν γίνονται όλα να μπουν σε μια έκθεση πρωτοβουλία. Οπότε καλό είναι να συγκεντρωθούμε, να δούμε πού πιέζουν τα προβλήματα. Βεβαίω, εμένα με ενδιαφέρει η αηφορία στον τομέα αυτόν και το πρόβλημα της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ξέρω από τον τομέα των βιολογικών προϊόντων που υπάρχουν πολλά προβλήματα διαφάνειας. Πού είναι αυτές οι δυσκολίες, ειδικά στο διασυνοριακό εμπόριο. Τα ξέρω λοιπόν κάπως ήδη στην πράξη και νομίζω αναφέρατε τα σημαντικότερα ζητήματα, αλλά πρέπει να δούμε κομμάτι-κομμάτι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και να αποκαταστήσουμε επίσης και μια επαφή με τις εκθέσεις που έχουμε κάνει ήδη, όπως αυτή για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή την έκθεση Fox για τα τρόφιμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα υπάρξει αυτή η σύνδεση για να μην κάνουμε δύο φορές τα ίδια. Επίσης κάτι το οποίο μου λένε από διάφοροι εκπρόσωποι δήμων τι συμβαίνει λοιπόν με τη γύρανση του πληθυσμού κατοικούνται όλο και πιο αραιά οι περιοχές της υπαίθρου και μετά τίθεται το ερώτημα μήπως ε, όλα αυτά γίνουν μια δημόσια υπηρεσία γιατί δεν είναι αρκετά επικερδή πλέον για τις επιχειρήσεις. Ο εφοδιασμός δηλαδή θα πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα λοιπόν, αλλά εμείς ως Επιτροπή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να επικεντρωθούμε σε κάνα δύο πράγματα και τα υπόλοιπα αργότερα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολύ περιεκτική ανάλυση που μας έκανε, επιμένοντας στα πιο σημαντικά θέματα και απαριθμώντας και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το εμπόριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως είπε σωστά εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λιανικό εμπόριο προσφέρει δουλειά σε πολλούς. Οπότε θα πρέπει στην πρότασή, μου, στην πρότασή μας να σεβαστούμε προϊόντα από όλες τις χώρες μέλη. Γιατί δεν θα πρέπει ένα μικρό αριθμό προϊόντων μόνο να κυκλοφορεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να υποστηρίξουμε και την τοπική γεωργία και του ντόπιου παραγωγού. Περιμένω να δω τι προσέγγιση θα θετήσει η συγγήτρια στο θέμα αυτό. Πάντως εμείς είμαστε έτοιμοι για συνεργασία καθ' τη διάρκεια των συζητήσεων. Και εγώ έχω κάποια σχόλια. γιατί είμαι σκιώδης της ομάδας μου για το θέμα αυτό. Καταρχήν συμφωνώ με όσους επισήμαναν ότι θα πρέπει οι σκιώδεις ε, μαζί με την εισηγητήρια να συζητήσουν το θέμα του πεδίου εφαρμογής ε, της έκθεσης αυτής για να μην ε, μπούμε στα χωράφια άλλων επιτροπών, αλλά να τους ζητήσουμε την γνωμοδότησή τους. Για παράδειγμα, από την Επιτροπή Γεωργίας που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η Γενική Διεύθυνση ε, Γεωργίας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων. Και είναι σωστό και αυτό που μου είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία σε ό,τι αφορά την πρόθεση των τόπιων παραγωγών και των προϊόντων που, έχουν, που μεταποιούνται και κυκλοφορούν πανευρωπαϊκά. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις, γιατί ήδη είχαμε ψηφίσει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την οποία καταθέσαμε και γνωμοδότηση. θα πρέπει να γίνει επικάλυψη με την έκθεση αυτή. Αυτό που με εντυπωσία στην παρουσίαση, ίσως όχι στην έκθεση, είναι ότι μιλάτε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το βασικό πρόβλημα όμως έγκυται κατά τη γνώμη μου στο ότι το δίκτυο αλυσίδες εφοδιασμού υπάρχουν προβλήματα και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αυτό είναι κάπως περίεργος. μιλήσατε για θέμητες εμπορικές πρακτικές, αλλά νομίζω ότι εδώ υπήρχε μια σύγχυση. Η νομοθεσία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές αφορά για τις ε, α, μεταξύ καταναλωτών. Ενώ εσείς μιλήσατε για στρέβλωση ανταγωνισμού μάλλον, για πρακτικές ε, αθέμητου ανταγωνισμού. Σε πολλούς α, ε, τομείς που εξετάσαμε, για παράδειγμα και για τα αυτοκίνητα, οι τοπικοί, εθνικοί περιορισμοί θεωρούνται ως σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εσείς είπατε ότι και οι ανέμποροι που θέλουν να αγοράσουν χονδρικά εμπόρια σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων δεν μπορούν να το κάνουν μερικές φορές, δεν μπορούν να αγοράσουν προϊόντα που φέρουν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού. Αλλά τώρα έχουμε και το scoreboard της αγοράς των καταναλωτών που κάνει μια αξιολόγηση της, κατάστασης και δείχνει πολύ σημαντικές διαφορές στις τιμές των προϊόντων μεταξύ των διαφόρων χωρών που δεν εξηγούνται από μια εύρυθμη λειτουργία αγοράς. Θα ήθελα αυτό το θέμα του ανταγωνισμού να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη και να μας καθησυχάσετε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς που έχουμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων, η δυνατότητα χονδρικής αγοράς και τη δυνατότητα που έχουν οι λιανέμποροι, ηλεκτρονικά δηλαδή να αγοράσουν χονδρικά, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το άνοιγμα της αλυσίδας εφοδιασμού. Νομίζω ότι αυτό δεν το καλύψατε παρκώς ε, στην παρουσίαση που μας κάνετε και θα ήθελα να το αναπτύξετε αν γίνεται αργότερα. Επίσης, ό,τι αφορά την ε, ίδια τη διάρθρωση του λιανικού εμπορίου και τις διαφορές ε, μεγέθους που παρατηρούνται. Σε πολλές περιπτώσεις εκφράστηκαν ανησυχίες για τις εξουσίες των μεγάλων λιανεμπόρων σε σχέση με τους μικροεμπόρους. Αυτά τα θέματα είναι σημαντικά για τον τοπικό προγραμματισμό. Και είπατε ότι αναπόκειται σε διακριτική ευχαίρεια αυτές οι προδιαγραφές προγραμματισμού. Θα πρέπει οι αρχές ανταγωνισμού να εξασφαλίζουν μια σωστή ισορροπία δυνάμεων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Και μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ζητήθηκε χαλάρωση των ε, προδιαγραφών προγραμματισμού για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ε, λιανεμπόρων. Δημιουργήθηκε ένταση όμως γιατί οι καταναλωτές μάλλον ήταν κατά. Πάντως ε, η αγοραστική δύναμη και οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι μεγαλέμποροι είναι θέμα αρκετά ανησυχητικό. Χθες ακούσαμε μία πληροφορία, ήταν και ο κύριος Αλντεμόζε, δεν θυμάμαι ποιος άλλος από την Επιτροπή, αλλά και ο κύριος Λούκεργαρτ, Ακούσαμε μια πολύ σημαντική παρουσίαση για την εφαρμογή του πακέτου και τις οδηγίες για τα προϊόντα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η ανοιχτή διακλαδική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είχαμε μια πολύ σημαντική μελέτη από έναν κατασκευαστή παιχνιδιών για προβλήματα ασυνεπούς εφαρμογής ή ελαττωματικής εφαρμογής των προδιαγραφών ε, για τα προϊόντα. Και το πρόβλημα είπε δεν είναι τόσο ότι οι κυβερνήσεις ή οι αρχές πιστοποίησης είναι περιοριστικές. Οι μεγαλέμποροι ζητούσαν έλεγχο των προϊόντων με βάση τις προδιαγραφές. Οπότε αν στέλναμε ένα προϊόν σε γερμανικά σούπερ μάρκετ θα ζητούσαν από εκεί επιπλέον ελέγχους αυτός ο κατασκευαστής ε, είχε έδρα την Ολλανδία και είπε ότι έλεγχος έγινε με βάση τις Ολλανδικές προδιαγραφές. Γιατί να μου τον έλεγχο με τις γερμανικές προδιαγραφές. Αλλά μερικοί ε, μεγαλέμποροι ελληνικού εμπορίου έχουν υπερβολικές ε, εξουσίες και ασκούν τεράστιες πιέσεις στο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις προσπάθειες της Γενικής Αστιεύθυνσης. Νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε εμείς να, αλλά και εσείς. Αλλά πουθενά στην έκθεσή σας δεν ε, αναφέρθηκε αυτό το θέμα. Μιλήσατε για τις προδιαγραφές που εφαρμόζουν οι λιανέμποροι και ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των κανόνων αυτών. Αλλά δεν είναι θέμα κανόνων, ε, είναι μάλλον θέμα θέμη των εμπορικών πρακτικών. Αλλά είναι αθέμητες οι πρακτικές όχι απέναντι στον καταναλωτή, αλλά απέναντι σε άλλες επιχειρήσεις. Και το γεγονός της χρήσης της αλυσίδας εφοδιασμού από ορισμένου λιανεμπόρους και η απέτηση που έχουν για υψηλότερες προδιαγραφές που ουσιαστικά αποθαρρύνουν την ε, είσοδο στην αγορά και πώς δημιουργούν έτσι εμπορικούς φαραγμούς, αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να βρεθούν στην καρδιά της έκθεσής σας και των προσπαθειών μας. Δεν είμαι βέβαιος ότι ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό όπως θα έπρεπε. Δεν νομίζω ότι του δώσατε τη δέουσα σημασία. Οπότε, χάρη στην ενεργό συμμετοχή της κυρίας Κοράτσα Μπίλ, που είναι συγκήτρια και συμμερίζεται τις απόψεις για το θέμα αυτό, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε σε αυτό το σημείο και την έκθεση επιτροπή. Ένα σχόλιο για τη Γερμανία. Το γνωρίζω το πρόβλημα. Το συζητήσαμε και για την οδηγία για τα παιχνίδια. Αν έχουμε αν είχαμε το third party certification, την πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο μέρος, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Ε, ίσως πρέπει να ξαναθέσουμε εδώ το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Άλλος κανείς. Ο κύριος Αμπάντ ήρθε για το επόμενο θέμα. Θα δώσω ξανά το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Περζεβά, για να απολογηθεί, μάλλον να υπερασπίσει τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες που του εξακόντισε και φυσικά και στην εισηγήτρια. Έχεις το λόγο, Ζαν, να μας πεις τη γνώμη έχεις και θα επανέλθουμε στην κυρία Κορατσαμπίλ και το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως, ε, σας ευχαριστώ για τα επικοδομητικά σχόλια και ευχαριστώ και για τα ωραία σχόλια. Υπάρχουν όμως και κάποια ερωτήματα και πριν αναφερθώ στο τελευταίο σημείο, το οποίο έθιξε και είναι πολύ σημαντικό, να πω το εξή. Σε απάντηση στα λεγόμενα της κυρίας Στήλε, νομίζω ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι, σημαντικ... είναι πολύ ε, σημαντικό. Εσείς το αναφέρατε ε, και εάν μπορεί κανείς να δώσει, να δώσει μεγαλύτερη δύναμη ε, στο τελικό χρήστη, έτσι ώστε να ξέρει ότι ας πούμε το ΑΒΓ μαγαζί έχει ε, θεσπίσει ήδη τις αρχές ποιότητας που αναφέρατε προηγουμένως, τότε η επιλογή του θα είναι πολύ πιο συνειδητή. Αλλά οι πληροφορίες που φτάνουν στον καταναλωτή είναι πολύ λίγες. Από την άλλη πλευρά, απ την άλλη πλευρά μιλώντας με τους λιανοπολιτές, ε, ξέρουν ότι όταν βάλουν, ε, εντάξουν στο δυναμικό τους ε, κάποια προγράμματα ποιοτικά κτλ, τα λεφτά τους τα παίρνουν πίσω ανταποκρίνονται οι καταναλωτές. Τώρα, Ε, υπάρχει μια, ένα μεγάλο πρόβλημα ε, το οποίο ονομάζουμε γενικά false return, ε, δηλαδή ψεύτικες επιστροφές, όπου ας πούμε ένας άνθρωπος σαν εμένα που δεν ξέρει καθόλου από τεχνολογία, αγοράζει μπαταρίες, τις χρησιμοποιεί λάθος, τις βάζει λάθος, πηγαίνει στο μαγαζί, λέω δεν λειτουργεί το μηχάνημα αυτό και δεν μπαίνει καν στον κόπο να το κοιτάξει λίγο και λέει καλά καλά εντάξει, ε, στο παίρνω και σου δίνω ένα άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ε, λυθούν. Πρέπει κάποιος να τα κάνει και βεβαίως θα θέλαμε να, να μάθουμε στους Λιανοπολιτές να τα κάνουν. Επίσης, το σημαντικό ζήτημα της βίας ε, στον χώρο εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμφωνούν ε, επί ενός κώδικα συμπεριφοράς για τον τομέα αυτό και επίσης μια συμφωνία και για το Eurocommerce και ε, ήδη, ασχολείται ένας φορέας με το θέμα αυτό. και επομένως ε, μπορούμε να γνωστοποιήσουμε ε, γενικότερα και αυτό που κάνει το Κοινοβούλιο και την εργασία άλλων φορέων. Τώρα όσον αφορά στον αντίκτυπο της ε, ύφεση, ε, κυρίως όσον αφορά τον σχεδιασμό. Ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κανόνες, συμφωνίες, κώδικες στα κράτη-μέλη που διέπουν τις συμβάσεις. Σε ορισμένες χώρες μέλη υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Αναγνωρίζουν ότι το λιανεμπόριο δεν μπορεί να έχει μεγάλη μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή ένα μεγάλο μαγαζί μπορεί να ε, πάει σε έναν άλλο δρόμο αρκετά μακρύτερα γιατί ε, το ενίκιο είναι πάρα πολύ ψηλό. Ένα μικρό μαγαζί δεν μπορεί να το κάνει γιατί θα χάσει όλη του την πελατεία. Θα πρέπει υπάρχουν κάποιες ε, χώρες οι οποίες ήδη έχουν εντάξει κάποια επιπλέον στοιχεία ε, στην ε, ευελιξία του λιανικού εμπορίου και επομένως εκεί μπορεί να έχουν κλείσει λιγότερα μαγαζιά ή να έχουν μετακινηθεί ε, η μικρή, το μικρό λιανεμπόριο. η αηφορία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Οπωσδήποτε το λιανικό εμπόριο καταβάλει προσπάθειες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν, ε, δεν απάντησα σε όλα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Όσον αφορά τις επικρίσεις, ναι, πιστεύω ότι το θέμα της... Το θέμα της αλυσίδας εφοδιασμού είναι όντως ε, κρίσιμο σημείο. Είναι γεγονός ότι πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, υπάρχουν προβλήματα, αλλά το πρόβλημα στην ουσία είναι διτό. Έχετε δίκιο ότι δεν μιλάμε εδώ για στρέβλωση των κανόνων ε, του ανταγωνισμού του εμπορίου. Μιλάμε για σχέσεις, για, για ε, εμπορικές πρακτικές. Μιλάμε για επιχειρήσεις. Μιλάμε επίσης για την δύναμη του, αγοραστή. Και επομένως μπορούμε να βάλουμε στις συμβάσεις τέτοια, ε, τέτοιες, τέτοιους όρους που ε, θα είναι οικονομικά δυσβάστακτο το βάρος μιας αλλαγής ε, πολιτικής. Δηλαδή, ε, αυτό είναι γεγονός ότι στο λιανικό εμπόριο είναι σημαντικό να έχει κανείς και συγκεκριμένες μάρκες, ας πούμε, μέσα στο μαγαζί του. Πρέπει να διευκολύνουμε την διαδικασία αυτή και σε πολλές περιπτώσεις εάν αρχίζει μια διαδικασία, αν αρχίσει κάπου μια διαδικασία whistleblowing μπορεί να έχει πολύ αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα ε, μαγαζί, σε ένα μικρό μαγαζί και προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε κάποιο σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί τελικά να έχουν πολύ κακό αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο. Ε, γενικότερα το θέμα δεν είναι μονάχα εάν υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος να καλύπτει ε, αυτή την λειτουργία whistleblowing. Ε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής του νόμου. από πλευράς εσωτερικής αγοράς οδηγούμεθα στο πρόβλημα το οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, τη διαφορά τιμών. Υπάρχουν αντικειμενικές ε, διαφορές, ε, μάλλον αντικειμενικά στοιχεία που οδηγούν σε διαφορά ε, τιμών. Αλλά τελικά υπάρχει και μία διαφορετική κίνηση σε σχέση με το ΑΕΠ. Θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι σε μία χώρα με ψηλό ΑΕΠ θα είναι ψηλές οι τιμές. Αλλά αυτό δεν ισχύει τελικά στην πραγματικότητα. Στις νέες χώρες μέλη βλέπουμε ότι η τιμή των προϊόντων συνήθως τίνει να είναι ψηλότερη. Ενδεχομένως αυτό οφείλεται ε, στην ε, ε, κακή διανομή, κακό σύστημα διανομής, κακή οργάνωση αλυσίδας εφοδιασμού. Αλλά πολύ συχνά έχουμε ανακαλύψει ότι αυτές οι υψηλές τιμές οφείλονται στα υψηλά ενίκια ή στην υψηλή αξία της ιδιοκτησίας. Επομένως είναι περίπλοκο όλο αυτό το σύστημα, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, είναι γεγονός. Μπορούμε να βρούμε τα επιμέρους προβλήματα, αλλά ε, γενικώ συμφωνώ ότι ειδικά για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είτε πρόκειται για λιανικό εμπόριο, είτε πρόκειται για μικρή εταιρεία μεταποίησης. Αναφερθήκατε και στο παράδειγμα των παιχνιδιών. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της αξιοπιστίας του λιανέμπορου, δηλαδή αυτό που αναφέρατε εσείς ως διαχείριση κινδύνου. Όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και ε, οι φορείς επαλήθευσης και ελέγχων ε, θα ε, ζητήσουν και πληροφορίες περισσότερες όταν, και από τους λιανέμπορους όταν μιλάμε για, κυρίως για προϊόντα τα οποία δεν είναι εθνικής παραγωγής. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και ένα πρόβλημα αξιοπιστίας τη πιστοποίηση και του ελέγχου γιατί θα πρέπει να σεβαστούμε τελικά και να πιστέψουμε τον έλεγχο που έχει γίνει σε μια άλλη χώρα ε, όταν ε, έχουμε εισαγωγή αυτών των παιχνιδιών. Και δεν μπορεί κανείς να δώσει μονάχα οικονομική εξήγηση στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα τέτοιου είδους. Τέλος, ζητώ συγγνώμη που δεν ε, αναφέρθηκα ε, στην ε, επιτροπή σας ως ε, του νου που κρυβόταν πίσω από την δημιουργία της νέας αγοράς, αλλά ναι, γνωρίζω την έκθεση του συναδέλφου σας στην οποία αναφέρατε και οπωσδήποτε αυτό θα μεταφερθεί στους συναδέλφους και δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τζον που ως συνήθως βεβαίως ε, είσαι στην Επιτροπή μας και ασχολείσαι με αυτές τις επικοδομητικέ προτάσεις, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ πέρα και νομίζω πως ε, είναι ζητήματα που μας έχουν ήδη απασχολήσει, έχουν ήδη αυτά τα οποία είπε η κυρία Σχάλδεμοζα για, Σχαλδεμόζα για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και όταν η κυρία Build, Κόρατσα build, θα συνδυάσει όλα αυτά, θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να τον λόγο για να μας πει τα των διαδικασιών και του μέλλοντος. Ευχαριστώ Μάλκομ. Μετά από την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση με τους κοιόδες ηγητές είχα την αίσθηση πως θα συνεργαστούμε καλά και σας ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια. Και να σας βοηθούν να δούμε το πεδίο εφαρμογής. Τρία πράγματα πρώτα απ' όλα. Πρέπει να δούμε το πεδίο εφαρμογής και το πώς θα το περιορίσουμε, αλλιώς δεν θα έχουμε σοβαρά και εις βάθος αποτελέσματα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, δηλαδή μπορούν να γίνουν σε κοινωτικό επίπεδο. Πολλά προβλήματα σχετίζονται με το ωράριο των καταστημάτων, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Πρέπει να δούμε πού θα έχουμε κοινού κανόνες και που αυτό θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χωροταξία που αναφέρατε. Η χωροταξία είναι πολύ σημαντικό η πολεδομία, αλλά συχνά γίνεται στο επίπεδο του Δήμου. Οπότε δεν νομίζω να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς αυτό. Σας ευχαριστώ επίσης ε, που το αναφέρατε αυτό, Μάικλ. Να σας υπενθυμίσω πως και εγώ είμαι φονταμενταλίστρια της εσωτερικής αγοράς. Πιστεύω στην εσωτερική αγορά. Και πράγματι ο τομέας λιανική είναι πυλώνας τη εσωτερική αγορά. Το να μην έχουμε κατακαιρματισμό είναι κάτι το τοθικό και για τους καταναλωτέ και για τις επιχειρήσεις. Και όπου είναι δυνατόν, εγώ είμαι υπέρ τη εναρμόνιση. Εγώ ίδρυσα και είχα μια μικρή εταιρεία, μιας, ε, μια μικρή εταιρεία τροφίμων, οπότε δεν χρειάζεται να πείστε εμένα Απλά θέλω να ελέγξω τα συναισθήματά μου, γιατί δεν θέλω τώρα να γίνει τελείω ιδεολογικό το ζήτημα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάντω ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές εταιρείε στην Ευρώπη, την κυρίαρχη θέση των μεγάλων αλυσίδων. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο πρακτικό, ρεαλιστικό και λογικό. Ευχαριστώ. Και αναμένω βέβαια συνεργασία με του συναδέλφου. Well, thank you very much. Uh, Well, I think as far as the timetable is is concerned, that, that yeah. Well, timetable. So, may I, Well, can I, I have say, the floor? I you may want to discuss. Well, you can talk about it if you like, but if we're going to have a... Ναι, κοιτάξτε, αν είναι να γίνει ακρόαση, ε, μπορεί να αλλάξει το, το χρονοδιάγραμμα. Οπότε καλό είναι ίσως να αφήσουμε τη συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, τι θέμε να κάνουμε. Αυτό προτείνω εγώ. Ναι, Συγγνώμη, να, να απαντήσω λίγο. Εγώ ε, ζήτησα ήδη μια κρόαση, δεν το ανέφερα γιατί είναι απόφαση που θα λάβουν οι συντονιστέν. Και ρώτησε τη γραμματεία μπορούμε να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε περισσότερο χρόνο για κρόαση και διαβουλεύσει. Οπότε οπωσδήποτε συμφωνώ, αναμένουμε προτάσεις. Θα είναι του χρόνου, δεν θα τελειώσουμε φέτος, αυτό προτείνω εγώ. Ναι, συμφωνώ και ειδικά ο νόμος περί εσωτερικής αγοράς θα έρθει κάποια στιγμή μέσα Οκτωβρίου, οπότε δεν νομίζω πως έχει νόημα. Ε, καλό είναι να γράψει την εκθεσή αφού υπάρξει ένα εργαστήριο, μια ακρόαση. Ε, οπότε αναμένουμε το έργο σας το οποίο οπωσδήποτε θα είναι με ενθουσιασμό. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας για την έκθεσή τους για μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης που νομίζω Σας παρακαλώ όσοι φεύγουν αν θέλουν έτσι λίγο με ησυχία κύριος Κρότσμαν θα μας εξηγήσει λίγο βέβαια τα πράγματα. Αυτό ήταν βασικό μέρος της Ατζέντα 2020 και νομίζω πως αναμένουμε ένα έγγραφο από την Κομισιόν που θα μας τα εξηγήσει εδώ πέρα αυτά τα πράγματα γιατί εγώ κάτι είχα δει κάποιος μου έδωσε κάτι κάπου Αναμένουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή Βιομηχανία και ο κύριο Κρότσμαν είναι ο εισηγητή και είμαι σίγουρο πω είναι πολύ έτσι χωμένος μας στο σύστημα και θα μας το πει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Μια βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη είναι κάτι το πολύ σημαντικό και διαπιστώνουμε πόσο συνεισφέρει η βιομηχανία στο ΑΕΠ αν το δούμε αυτό, διαπιστώνουμε πως εντός της Ευρώπης έχουμε πολύ διαφορετικές δομές. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, μιλάμε για ένα 25% συνεισφορά στο ΑΕΠ. Αν πάρετε την Αγγλία, μιλάμε για κάτι λιγότερο από 15%. Οπότε, πρέπει να δούμε κατά πόσον ενδιαφέρονται τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν πως είναι προς το συμφέρον τους να προωθήσουν μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Το είδαμε π.χ. κατά τη διάρκεια της ε, οικονομικής κρίσης πως η Γερμανία είχε αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και αύξηση ε, κατά 3% του ΑΕΠ και αποτέλεσε την αγρομηχανή τη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να σκεφτούν πώς πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για να ενισχύσουν τη βιομηχανική τους παραγωγή. Βεβαίω τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν στο πώς θα κατευθύνουν την ε, πολιτική τους για να έχουν μια ανταγωνιστική βιομηχανία. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, δεν υπάρχει μόνο η Ευρώπη. Οπότε, στον καιρό της παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει η βιομηχανική πολιτική να διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι ένας κινητήρας, να έχουμε ευκαιρίες εντός της Ευρώπης και να παράγουμε τα προϊόντα μας παγκοσμίω. Και αυτό το οποίο είπε ο Λάγγεν είναι μια πάρα πολύ καλή βάση και νομίζω μπορούμε να συμπληρώσουμε διάφορα πράγματα ή να δούμε εάν θα κάνουμε κάποιες προτάσεις εσωτερικής αγοράς. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να δώσω βάρος στις προτάσεις εσωτερικής αγοράς που είναι βέβαια η Επιτροπή μας αλλά δεν νομίζω θα είναι άσχημο να δουμε εαν θα κανουμε καποιες προτασεις εσωτερικης αγορας αυτο το οποιο θελω να κανω ειναι να δωσω βαρος στις προτασεις εσωτερικης αγορας που ειναι βεβαιος η επιτροπη μας αλλα δεν νομιζω θα ειναι ασχημο να υπαρξει και καμία συμπλήρωση σε αυτά τα οποία υπέβαλε ο συνάδελφος του Επιτροπής Μηχανής. Η πρόταση καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα, καινοτομία, πολιτική έρευνας, αλλά βλέπουμε πως η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για στήριξη της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη. Στην γνωμοδότησή μου αναφέρω πως ε, σημαντικό είναι να υπάρχει μια, ένα πλαίσιο φορολόγησης της βιομηχανίας, δηλαδή να αποφύγουμε τις ακραίες καταστάσεις που είχαμε, όπως στον τομέα τον χρηματοπιστωτικό, αλλά πρέπει να αφήσουμε ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις ε, ένα χώρο έλιγμων για να βρεθεί καλύτερη λύση μέσω του ανταγωνισμού γι' αυτό. Η δημιουργία του σωστού πλαισίου, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, π.χ. η κατάργηση της γραφειοκρατίας είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η ολοκλήρωση λοιπόν της εσωτερικής αγοράς σημαίνει πως θα πρέπει να έχουμε αναλόγες εθνικές στρατηγικές. Η έκθεση Μόντι έδειξε πως πρέπει να υπάρξει δράση και τώρα η Κομισιόν στο πλαίσιο της αγώνησης εσωτερικής αγοράς εξετάζει τον νόμο περί εσωτερικής αγοράς για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη και αποτελεσματικότερη εναρμόνιση. Θεωρούμε λοιπόν πως μια οδηγία εδώ πέρα έχει πάρα πολύ καλό δυναμικό. Επίσης ζητάμε από τα κράτη-μέλη να παίξουν έναν ενεργητικό ρόλο στη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς και οι αριθμικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνεχώς διαπιστώνουμε πως κανόνες, οδηγίες, ε, κανονισμοί εκδίδονται, αλλά βλέπετε πως το πρόβλημα μετά είναι στην εφαρμογή στα κράτη-μέλη, όπως έδειξε και η οδηγία των υπηρεσιών πρωτοβουλία νομίζω για την ε, απλοποίηση της νομοθεσίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας έχει ήδη επιφέρει αποτελέσματα, αλλά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα να φύγουν οι αντιφατικές διατάξεις. Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία και να επεκταθεί. Επίσης, σωστή νομοθεσία θα πρέπει να γίνονται οι σωστές εκτιμήσεις αντικτύπου στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και να γίνουν πιο στηματικές. Ακριβώς όσον αφορά δε και το μέλλον της ε, τυποποίησης για την οποία μόλις ψηφίσαμε, αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ενίσχυση των εθνικών εδώ πέρα διατάξεων. Επίσης για τους εθνικούς διαγωνισμούς θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να είναι ανοιχτοί και πιο απλοί οι κανόνες, να υπάρχουν ελάχιστες ε, κοινοτικές προδιαγραφές κριτήρια. Επίσης καινοτομία για το περιβάλλον τα οποία θα πρέπει να περιέχονται στους δημόσιους διαγωνισμούς. Η βιομηχανία ζητάει επίσης αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και εκτός εσωτερικής αγοράς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα συνεισφέρει λοιπόν εδώ πέρα μια τυχόν συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Επίσης είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να μην έχει η ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία απαιτήσει οι οποίες δεν υπάρχουν από τους ανταγωνιστές τους. Αυτό το λέμε πάντα όταν μιλάμε για το εμπόριο εκπομπών. Εάν κάνουμε εμείς κάτι τέτοιο, ε, οι άλλοι δεν το κάνουν, οπότε τι κάνουμε, επιβαρύνουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα που πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην σημασία τεχνολογιών κλειδιών. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να δώσουμε βάρος στο ότι θα πρέπει να υπάρχει κρατική ενισχύση η οποία όμως θα συμμορφώνεται πλήρως με τα του ανταγωνισμού και οι επενδύσεις θα πρέπει βεβαίως να είναι δουλειά της βιομηχανίας, θα πρέπει το κράτος να φροντίζει για την αποδοχή νέων τεχνολογιών, όπως παραδείγματο χάρη η βιοτεχνολογία. Και όταν αυτό βεβαίως βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε. Η βιομηχανική πολιτική είναι σημαντική Όσα κράτη-μέλη θεωρούν πως μπορούν να ζήσουν μόνο με υπηρεσίες, ε, έχουν τώρα καταστροφικές εξελίξεις, τις είδαμε στον τομέα των χρηματοπιστωτικό και η άποψή μου, επειδή ανέφερα και την ε, Αγγλία, που έχει λιγότερο από 15% συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, υπάρχουν και εκεί πέρα να αναζωογονηθεί η βιομηχανική παραγωγή για να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Και αν δει κανεί τη Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία ήταν το βιομηχανικό κράτος ε, τους περασμένες ε, δεκαετίες. Οπότε θα πρέπει να δώσει μία όθηση. Είμαστε πρώτο πόροι στην Ευρώπη όσον αφορά την ιατρική τεχνολογία, σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Καμιά φορά το θέμα είναι η εφαρμογή, δηλαδή κάνουμε εμείς την ανακάλυψη και την παραγωγή την κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι. Εκεί πέρα μπορούμε να συνεισφέρουμε. Τέλος, κάποιες παρατηρήσεις για το χρονοδιάγραμμα που θα θέλετε να το ξέρετε. 11 Οκτωβρίου παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης προθεσμία για τροπολογίες 13 Οκτωβρίου 12 η ώρα και ψηφοφορία 18 Νοεμβρίου. Αυτά προτείνω εγώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ah, well, thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Κρόιτσμαν. Πολύ ενημερωτική αυτή η παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάνφρετ Μπέρκμαν από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ένα δεκάλεπτο μας έχει μείνει μόνο, αλλά θα του δώσω το λόγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κρόιτσμαν, αν περιμένουμε όντως την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν έχουμε λάβει ακόμη την ανακοίνωση αυτή για την βιομηχανική πολιτική την εποχή παγκοσμιοποίησης. Είναι η δεύτερη έκθεση που αφορά τη στρατηγική για το 2020. Τι είπατε για τον κύριο Λάγγεν, ότι θα ολοκληρώσει την έκθεσή του πριν δημοσιευθεί αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θα την περιμένει δεν ξέρω, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων θα μπορεί να μας πει πότε σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει αυτή την ανακοίνωση για να εξετάσουμε και το χρονοδιάγραμμά μας και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έγκριση της ανακοίνωσης προβλέπεται για τις 27 Οκτωβρίου. και η πρωτοβουλία για την κοινοτομία θα εγκριθεί στις 26 ε, Οκτωβρίου. Οπότε και στις 19 Οκτωβρίου το Single Market Act, αυτή η πράξη για την ενιαία αγορά. Αυτό είναι ενδεικτικό με το χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζουμε θα το τηρήσουμε, εκτός και αν ε, ε, προκύψουν απρόβλεπτες δυσκολίες, αλλά το απέφχομαι. Αυτή την εντύπωση είχα και εγώ, λέει ο κ ότι αυτές ήταν οι προθεσμίες. Γι' αυτό πρότεινα και εγώ το χρονοδιάγραμμα που σας υπέβαλα. Ναι, αλλά η περισσότερο για τον ε, κύριο Λάγκεν της αρμόδιας κατουσίαν επιτροπής, της Ήτρε. Γιατί αν εμείς ε, το υποβάλλουμε για τις 13 ε, Οκτωβρίου, εκείνος θα εγκρίνει στην Ήτρε την έκθεση την, τον ίδιο καιρό με την δημοσίευση της ανακοίνωσης Επιτροπής. Δεν ξέρω πώς θέλει ο κύριος Λάγκερ να καθυστερήσει την έγκριση της έκθεσης για αρκετές εβδομάδες προκειμένου να λάβει στο μεταξύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μπορέσει να τη σχολιάσει. Αλλά αυτό καλύτερα να το δείτε εσείς μαζί με τον κύριο Λάγκερ γιατί είναι σε πολύ προχωρημένη φάση η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την περιμένουμε σχετικά σύντομα, οπότε Χρήσιμο ήταν να περιμένουμε την ανακοίνωση, να δούμε τι μορφή θα έχουν οι προτάσεις για να μπορέσουμε να τις σχολιάσουμε. Οπότε, αν παρατείνουμε το χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει ζήτημα. Καλά, στο αφήσουμε προς το παρόν, θα δούμε. Ζήτησαν το λόγο ο κύριος ε, Ματ, Κορέο Δεκάμπος, ο κύριος έφυγε στο μεταξύ. θα κάνω εγώ σύντομα σχόλια, θα ακούσουμε τον κύριο Μπέργκμαν και ελπίζω το 12.30 να προλάβουμε να τελειώσουμε. Ο κύριος Αμπάντ πρώτα. Ευχαριστώ. Για το χρονοδιάγραμμα και εγώ προτιμώ να περιμένουμε την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν υποβάλουμε την γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η βιομηχανική πολιτική είναι προτεραιότητα. Και εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για αρκετό καιρό είχαμε μια αντιπαλότητα της ε, βιομηχανικής πολιτικής και της εσωτερικής αγοράς. Τώρα έχουμε όμως και το Single Market Act, αλλά και τη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική που θα μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες για να ξανασυμφιλιώσουμε την εσωτερική αγορά με τη βιομηχανική πολιτική. Έχουμε και θέλουμε μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική που θα δημιουργεί ευκαιρίε για όλε τι επιχειρήσει και ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε. Θα πρέπει να δούμε τι επίπτωση έχει η βιομηχανική πολιτική στην εσωτερική αγορά και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ανανεώσουμε την πολιτική των κρατικών προμηθειών αφήνοντας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να καρποθούν ένα τμήμα του μεριδίου των ε, δημοσίων προμηθειών. Φυσικά, λαμβάνοντα υπόψη περιβαλλοντικέ ε, και κοινωνικέ επιταγέ, αλλά και την ανάγκη τη καινοτομία. Επίση, το θέμα τη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Να αποφευθεί ο κατακαιρματισμό των κεφαλαίων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις, τα δάνεια κινδύνου και να εμπλέξουμε όσο δυνατό περισσότερους ενδιαφερομένους ε, προωθώντας και συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Θα πρέπει επίση να προωθήσουμε και να δώσουμε ανάψματα στους πλέον καινοτόμους τομείς, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Εκτός από την εσωτερική όμως διάσταση της ε, εσωτερικής αγοράς, έχουμε και μια εξωτερική διάσταση. Θα πρέπει να διεκδικούμε αμοιβαιότητα και αντίστοιχα ωφέλη με αυτά των εταίρων μας. Και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η αμοιβαιότητα στην πρόσβαση σε επιχειρήσεις, γιατί οι ιαπωνικές αγορές έχουν 75% πρόσβαση στις δικές μας κρατικές προμήθειες, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν μόνο 35% πρόσβαση στις ιαπωνικές κρατικές προμήθειες. Επίσης θα πρέπει να καταλύσουμε τις παραποίησεις. Είναι σημαντική προτεραιότητα της βιομηχανικής πολιτικής να προσπίσουμε τις τεχνογνωσίες, την τεχνογνωσία της βιομηχανικής μας πολιτικής. Θα πρέπει να προωθήσουμε προγράμματα και σχέδια που θα ωφελούν και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και με πολύ δραστηριό τρόπο και επιθετικό να προωθήσουμε μια βιομηχανική πολιτική που θα συνάδει με τις απαιτήσει και τις εσωτερικές αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπάτ. Πολύ χρήσιμα και εύστοχα τα σχόλιά σας και συμφωνώ ε, μαζί σας θα πρέπει να συνεργαστούμε και να τονίσουμε και την εξωτερική διάσταση. Εγώ είμαι μέλο και τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Ιαπωνία και εκεί αναφέραμε αυτό το θέμα της ε, πρόσβασης στις ε, δημόσιε αγορές και κρατικές προμήθειες. Κύριε Κάμπος, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Μπέργμαν και τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη σωστής διαχείρισης του χρονοδιαγράμματος και σωστού συγχρονισμού. Γιατί όσο ευρηματικοί και αν είμαστε και φάνταστοι, καλύτερα να αξιοποιήσουμε και το έργο και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσοχή λοιπόν στο χρονοδιάγραμμα, σωστό συγχρονισμός για να δρέψουμε όσο το δυνατό περισσότερους καρπούς από αυτή την συνεργασία. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον εισηγητή Κρόιτσμαν. Θα προσθέσουμε και κάποια νέα σημεία σίγουρα και θα εμπλουτίσουμε την έκθεση Λάγκε της Επιτροπής Βιομηχανίας. Συμφωνώ απόλυτα με την πολιτική σημασία που δίνουμε πια στη βιομηχανική πολιτική. Γιατί κάποια στιγμή ακούσαμε ότι είναι τελείως άχρηστη η βιομηχανική πολιτική. Είδαμε όμω τις διαφορέ μεταξύ του 25% της Γερμανίας και του 15% της Μεγάλης Βρετανίας και τι τεράστιες διαφορέ υπάρχουν. Είναι λοιπόν επιτακτική πλέον η ανάγκη της δημιουργίας μιας βιομηχανικής πολιτικής. Συμφωνούμε και με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη σημασία που θα διαδραματίσει η ενιαία εσωτερική αγορά στην ανάπτυξη μιας βιομηχανικής πολιτικής μέσω διαφάνειας των διαγωνισμών, θέσπισης σημαντικών προδιαγραφών. Μάλιστα θα έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση για αυτό το θέμα, άρα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και το καθεξής. Αλλά δεν μπορούμε να προτείνουμε μια βιομηχανική πολιτική που θα είναι παροχημένη. Ε, θα πρέπει να βρούμε τους ε, θύλακες, τα συγκριτικά ωφέλη. Το θέμα των νανοτεχνολογιών ή των ιατρικών τεχνολογιών είναι πολύ σημαντικά. Γιατί εκεί είμαστε προηγμένοι και εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Επίση, έχουμε πολύ περίπλοκα θέματα ενό προηγμένου συστήματος υγείας που δημιουργεί όλο και νέες ανάγκες. Και θα πρέπει να δούμε ταυτόχρονα τη βαριά βιομηχανία που εξάγει και απασχολεί πολύ εργατικό δυναμικό, όπως είναι η το αλλά να δούμε και την κατάσταση των βιομηχανιών ε, ε, καινοτόμων τομέων, ε, νης, θυλάκων, γιατί και αυτές δίνουν έφεση στην καινοτομία και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Συγχαίρω και τον εισηγητή για τα σχόλιά του, αλλά και τον κύριο Μπάτ για τα δικά του σχόλια που ήταν πολύ εύστοχα και τεκμηριωμένα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά ίσως ο Δόκτωρ Μπέργκμαν θα μπορούσε σε πολύ λίγο χρόνο να μας πει δύο λόγια. να εστιάσει στο ενδεχόμενο μελλοντικής, ε, της μελλοντικής ανακοίνωσης και μετά ο κύριος Κρόιτσμαν να ε, ολοκληρώσει και βεβαίως η Γραμματεία να μιλήσει με τον κύριο Λάγκεν για να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις διορίες. Δόκτωρ Κρόιτσμαν. Μπέργμαν, συγγνώμη. Βεβαίω είναι πολύ πρόημο για να ε, προβλέψει κανείς ποιες γενικές γραμμές θα εγκριθούν. Είναι σαφές ε, όμως ότι ο κύριος στόχος είναι να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιομηχανική βάση της Ευρώπης. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε, ε, να, ε, ε, είναι σαφής η τάση για εκδίωξη των βρώμικων ας πούμε βιομηχανιών και βελτίωση των συνθήκων. Επίσης, ευελπιστώ ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ε, θα αντλήσουν ιδέες ε, κοινέ και ότι ε, φαίνεται ότι και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν βλέπουν το θέμα υπό το φως και της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας. Έχω δει την, το προσχέδιο του κυρίου Λάγκεν και διαπιστώνει κανείς ότι γίνεται 30 φορές αναφορά στην ε, ε, βιωσιμότητα και την αηφορία και 10 φορές μονάχα στην ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αηφορία ε, χωρίς ανταγωνιστικότητα, ούτε ανταγωνιστικότητα χωρίς καινοτομία. Επομένως λοιπόν αυτά τα διάφορα στοιχεία δεν θα πρέπει να τα δούμε μεμονωμένα το καθένα, αλλά ε, σαν κοινά στοιχεία, μιας, σαν στοιχεία μιας κοινή προσπάθειας. Και παραπέμπω εδώ και στην ε, ανακοίνωση για την ενιαία αγορά και για την ε, ε, δυνατότητα αυτάρκειας εφοδιασμών. Νομίζω ότι ε, κανείς δεν πρέπει να βλέπει κάποια πρωτοβουλία ξέχωρα από άλλες υφιστάμενες. βλέποντας ε, και την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την πρόσφατη οικονομική κρίση, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ε, μια κοινή σκέψη καλή. Βεβαίως δεν αρκεί η ενδυνάμωση ενός μεμονωμένου στοιχείου. Ε, θα πρέπει να ε, δει κανεί όλα τα στοιχεία της αλυσίδας και επίσης μας ενδιαφέρει να μην υπάρξει μετατόπιση ή υποτίμηση κάποιων μεμονωμένων στοιχείων αυτής της αλυσίδας. Ένα δεύτερο μάθημα που μάθαμε από την ε, κρίση και που αναφέρεται στην ανακοίνωση είναι το θέμα των ε, μεμονωμένων ε, εθνικών και απομονωμένων εθνικών βιομηχανιών που φαίνεται να μην έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής πλέον. Λέμε ότι οι αξίες, οι αλυσίδες αξιών είναι σημαντικές ε, και αυτές οι αλυσίδες θα πρέπει να είναι σε εθνικό αλλά και σε διεθνικό επίπεδο. Και ε, θέλουμε ε, κατά αυτή την έννοια καλύτερη και δυνατότερη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και να ενδυναμώσουμε την ενιαία αγορά γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά στην Επιτροπή σας η ενιαία αγορά είναι ένα ε, σημαντικό προπύργιο απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο, απέναντι στα προβλήματα ε, και επομένως ε, θα πρέπει να δούμε και το θέμα των υποδομών και το θέμα της αναδιανομής και πολλά ζητήματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν από κοινού ε, πιο ε, έξυπνη, ε, πιο έξυπνος διακανονισμός, πιο έξυπνο ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας να βελτιωθεί. Και τέλος, όταν μιλάμε για εξωτερήκευση, όταν μιλάμε για προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι πολύ σημαντικό να καταβληθούν όλες οι ε, προσπάθειες έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος του επιχειρήν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι η δουλειά και της Επιτροπής σας και των λοιπόν θεσμικών οργάνων. διότι το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο και περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν καταβληθεί, εξεκολουθεί να είναι εξαιρετικά καταγερματισμένο. Επομένως, ε, ε, αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Ευχαριστώ. δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Λοιπόν, για να δούμε. Βλέπουμε εδώ πέρα ε, πως πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα έκθεση και δεν ξέρω, νομίζω οι συνάλφοι έχουν δίκιο. Πρέπει να ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα. Και χάρηκα ιδιαίτερα για το ότι αναφέρατε κάποια από τα σημεία αυτά και αυτό το οποίο είπε ο πριν. Και Κρότσμαν, έχετε να κάνετε άλλα σχόλια. Πριν ε, λήξει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκαν πάρα πολλά, αλλά πρέπει να πούμε πως έδειξαν οι σκιώδες ομιλητές πόσο σημαντική είναι η βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή η βιομηχανική πολιτική πρέπει να ενισχύει τη βιομηχανία. Χωρίς ε, ανταγωνιστική ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Το βλέπουμε αυτό. οι Αμερικανοί που ήταν τόσο υπερήφανοι για τις υπηρεσίες τώρα παραπονιούνται πως οι εξαγωγές στην Κίνα ή δεν ξέρω και εγώ που δεν ε, υπάρχουν. Οπότε οι υπηρεσίες θα υπάρχουν όταν υπάρχει και βιομηχανία. Οπότε νομίζω πως θα είναι καλή αυτή η έκθεση και πηγαίνουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Well, thank you uh, everybody very much for those contributions. Um... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω λοιπόν πως με την ευρία εντολή που έχει η Επιτροπή μας, το απόγευμα θα δούμε τις δραστηριότητες του κλάδου των υπηρεσιών. Όπως είπε βέβαια, ο κύριος Κρότσμαν, πρέπει να το δούμε αυτό από κοινού με τη βιομηχανία. Και η συνεδρίαση θα ξεκινήσει τρεις και μισή, όχι τρεις. Θα γίνει ένα εργαστήριο, μια παρουσίαση μια ενημέρωση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε ξανά εδώ ραντεβού 3 και μισή. Και αυτό είναι το μόνο θέμα στη μερίσια διάταξη του απογεύματο. Να υπενθυμίσω επίσης στου συντονιστές πως αύριο το πρωί στις 9.30, 9 συγγνώμη, συνεδριάζουμε και 10 και μισή, μια άλλη σημαντική ακρόαση κυρία κυρίας Μόζε για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία τη αγορά θα έχουμε και μία ενημέρωση από ειδικού. Ελπίζω να έρθετε λοιπόν. Κυρία Μόζε, θα προεδρεύει γιατί εγώ πρέπει να πάω στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα αύριο για να εκπροσωπήσω την Επιτροπή μας. Και να σας πω